No, yeah, but I mean, uh, <laughs> you can be a little bit late. <laughs> Okay. Eh, buenos días, vamos a Καλή σα ημέρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ε, ελπίζω να έχετε φέρει τις ε, κάρτες για τις ψηφοφορίες, ε, διότι θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες που βλέπονται για σήμερα. Ως πρώτο σημείο έχουμε την έγκριση της μισής διατάξεως. Να σας ανακοινώσω Πώς η κυρία Πατράου ζήτησε το σημείο 9 σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα στήριξης περαιτέρω με μεκροχρομές θαλάσσιας πολιτικής να εξεταστεί μετά από τις ε, ψηφοφορίες ε, διότι θα χρειαστεί να αναχωρήσει. Ως εκ τούτου, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα εξετάσουμε το σημείο 9 μετά από τις ψηφοφορίες και με τον τρόπο αυτό τροποποιούμε τη μέσα διάταξη αν φυσικά δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, και να σας ε, ανακοινώσω πως ε, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μεσής διατάξης, έγκριση των πρακτικων συνεδριάσεων 25-26 Ιανουαρίου του 2011 και 1 Φεβρουαρίου του 2011. Αν κατά τη διάρκεια συνεδρίαση σήμερα το δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, τότε θα θεωρηθούν σε εγκρίνονται. Το σημείο 3 δεν έχω να σας ε, κάνω καμία ανακοίνωση. Το σημείο 4 είναι η ψηφοφορία του πρώτου θέματος ε, σε ό,τι φορά τους κανόνες εισαγωγής από τη Γρυλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελευτικών προϊόντων, ζώντων, δίθυρων, μαλακίων κλπ. Εγώ είμαι η συγγήτρια Γνωρίζετε πως ε, το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε επανειλημμένος ε, και το μοναδικό πρόβλημα είναι η νομική βάση. Λάβαμε υπόψη της απόψεις της νομικής υπηρεσίας και της ε, νομικής επιτροπής που στήριζε τη τροποποίηση της νομικής βάσης και ως εκ τούτου οι τρεις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έχουν άμεση διασύνδεση με την νομική βάση διότι επιθυμούμε να την τροποποιήσουμε. Αν ε, δεν υπάρχουν ενστάσεις, ε, ξεκινάμε και ψηφίζουμε ομού τις τροπολογίες, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 ψήφισαν, 18 ψηφί, υπέρ, εγκρίθηκαν οι τροπολογίες Ορίστε, θέλετε το λόγο. Α, δεν έχετε την κάρτα σας. Ε, όλα τα περιπλέκουμε τα πράγματα, εντάξει. 20 οι ψήφοι λοιπόν, διότι δύο συνάδελφοι δεν έχουν την κάρτα τους. Ε, με τώρα το εντρομένη πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος, ε, αρχή ψηφοφορία, πέρα ψηφοφορίας. Και εδώ έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, 20 ψήφισαν, 20 ψήφι υπέρ. Και τώρα περνάμε στο ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίζουμε. Έληξη ψηφοφορία. Και εδώ ομοφωνία λοιπόν. Περνάμε τώρα το επόμενο θέμα πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Κάπουλα Σάντο, πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό αλληλευτικών δυνατοτήτων και χρηματική αντιπαροχή. Βλέπω για συμφωνία αλληλευτική συμπρέχει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κομορών. Ε, εδώ έχουμε την διαδικασία τη ε, σύμφωνη ε, νόμη και πρέπει λοιπόν να δεχθούμε την συμφωνία όπως πρότεινε ο κ. Κάπουλας. Θέλετε το λόγο κύριε Κάπουλα, όχι. Να ψηφίσουμε λοιπόν. την ε, έγκριση της ε, συμφωνίας, της συνένεση μάλλον, πέρα ψηφοφορίας. 20 οι ψηφίσαντες, 18 ψήφοι υπέρ και 2 κατά. Εγκρίθηκε λοιπόν. Και τώρα περνάμε στο ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 20 ψήφισαν, 18 ψήφι υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Δεκτή. Συγχαρητήρια κύριε Κάπουλα Σάντος. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μεσής διατάξεως. Πρόκειται για την ε, ε, απαλλαγή 2009 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου Αλίας. Συγητής είναι ο κύριος Γκάλαχερ. Θέλει να λάβει το, να το λόγο, όχι, ψηφίσουμε. Υπάρχει τροπολογία στην παράγραφο 3 της κυρία Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπερθμών 1. Έληξε η ψηφοφορία. 20 ψήφισαν, 20 ψήφοι υπέρ, και τώρα ψηφίζουμε στο, το σύνολο ε, του σχέδιου γνωμοδοτήσεως. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 ψήφισαν, 20 ψήφι υπέρ. Συγχαρητήρια κύριε Κάραχερ, δεκτή η νομοδότησή σας, τα συγχαρητήριά μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μισής διατάξεως. Πρόκειται για την έκθεση της κυρίας Πατράου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Γνωρίζετε πως ε, έγινε σε συνδυασμό με την Επιτροπή Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 50 και δίνω το λόγο στην κυρία Πατράου. Señora Πατράου, tiene usted la palabra. Έχετε το λόγο, κύριε Πατράου. Καλημέρα. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να ξεκινήσω. Περιμένω λίγο να ηρεμήσουμε στην αίθουσα. Ναι, ναι. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία γιατί περιμένει η κυρία Πατράου για να ξεκινήσει. Παρακαλώ ξεκινήστε εσείς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ να σας πω, θέλω να σας πω το εξή. Εγώ δεν ζήτησα να αλλάξει η μερική διάταξη. Η γραμματεία μου το ζήτησε. Εγώ δεν ε, παρουσίασα κανένα πρόβλημα. Δεν ήταν δίκη μου πρωτοβουλία δηλαδή αυτή η τροποποίηση της ημερησίας διάταξης. Σήμερα το θέμα που σας παρουσιάζω είναι η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα στήριξης περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Να υπενθυμίσω ότι το 2006 με την παρουσία από την Κομισιόν της Πράσινης Βίβλου για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που ξεκίνησε η δημιουργία αυτής της πολιτικής ε, Πρέπει να φτάσουν ε, το μέγιστο, να φτάσουμε στο μέγιστο της ε, εκμετάλλευσης της θάλασσας και αυτή η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική βασίζεται στο ότι μπορεί να έχει πολλές χρήσεις η θάλασσα και ακριβώς από εκεί προκύπτει και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Και όταν μιλάμε για αυτή την πολλαπλή χρήση, δεν μιλάμε μόνο για του παραδοσιακού τομεί που χρησιμοποιούν τη θάλασσα για τη θεμελιώδη δραστηριότητά του, όπω ε, η αλία και οι μεταφορέ, αλλά πιο πρόσφατα μιλάμε για δημιουργία αιωλικών ε, υπεράκτιων πάρκων, ε, επένδυση τεχνολογιών σε σχέση με την κλιματική ενέργεια, υδατοκαλλιέργεια υπεράκτια και πολλές άλλες πτυχές ε, που αποκαλούνται σήμερα βιοτεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίστηκε ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Είχαμε την παρουσίαση μια ανακοίνωση ε, μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Το έγγραφο αυτό προβλέπει δύο μεγάλες συνιστώσεις δράσης. Καταρχήν, τομεακές δράσεις ε, στον ε, τομέα της ενέργειας, των μεταφορών, της έρευνας, των επαγγελμάτων και των εξωτερικών σχέσεων, αλλά και ταυτόχρονα τη δημιουργία δομών διακυβέρνησης που μπορούν να εγγυθούν τις αντίστοιχες θαλάσσιες πολιτικές έτσι ώστε να υπάρχει διάρθρωση μεταξύ των πολιτικών αυτών. Και στο πλαίσιο αυτό Σήμερα βλέπουμε την Αλία. Η Αλία δεν μπορεί να βρίσκεται εκτό τη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Πρέπει να είναι εντό και πρέπει να έχει και ένα ρόλο παρεμβατικό σε αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αυτό μάλιστα γιατί αυτή θα είναι και μια πτυχή που θα προσδώσει ένα πλεονέκτημα στην Αλία. Γιατί ε, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής μπορούμε πράγματι να κερδίσουμε προβολή για την ιδιαιτερότητα του τομέα της Αλίας. Έτσι λοιπόν και πάντοτε έχοντας κατά νου ότι πρέπει να αναγνωριστούν και ιδιαιτερότητες της αλίας σε ό,τι αφορά τη χρήση της θάλασσας. Έχοντας λοιπόν έτσι τα πράγματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτό, πράγματι, προκύπτει συγκεκριμένη πρόταση κανονισμού που μας απασχολεί εδώ σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα για το θέμα αυτό θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο εξή αφού ζητήσαμε ενισχυμένη συνεργασία για να γίνουμε συνδεόμενη επιτροπή και να μην επιτρέψουμε να είναι επί η Επιτροπή Μεταφορών, η επί της ε, ουσίας αρμόδια Επιτροπή. Αυτό έχει θετικά αποτελέσματα και φυσικά αυτό μας ικανοποιεί όλους. Γνωρίζουμε ότι ήδη εδώ και πολύ καιρό Είχαμε συζητήσει η αναγκαιότητα της Επιτροπής Αλίας να έχει αυτό το καθεστώς της Συνδεδεμένης Επιτροπής και στις 10 Ιανουαρίου μας χορηγήθηκε αυτό το καθεστώς και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το έγγραφο αυτό και για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και για το ότι η Αλία σε αυτό το πλαίσιο τη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική διαδραματίζει ένα ρόλο ισότιμο με των μεταφορών, αλλά δημιουργείται και ένα σημαντικό προηγούμενο για το μέλλον σε σχέση με άλλα ζητήματα για τα οποία θέλουμε να έχουμε και πάλι αυτό το καθεστώς της Συνδεδεμένης Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, προτάσεις ε, τρόπολογιών στο βασικό κείμενο που παρουσιάστηκε, θα έλεγα ότι εδώ έχουμε τρεις κυρίες πτυχές. Ο ένας πρώτος στόχος από τη δική μου πλευρά ήταν να καταστήσω το έγγραφο πιο διαρθρωμένο, πιο ομοιογενές και γι' αυτό εδώ έχουμε πολλές ε, που ίσως φαίνεται υπερβολική εκ πρώτες ε, όψεως, όμως ε, πρόκειται πράγματι για αναδιοργάνωση του εγγράφου, αναδιάρθρωση του εγγράφου σύμφωνα με μια θεματική αλληλουχία. Αυτό συμβαίνει κυρίως στα άρθρα 2 και 3. Στα άρθρα 2 και 3, τα άρθρα αυτά είναι αναδιαρθρωμένα και ταυτόχρονα προσπάθησα να ενισχύσω και τους κύριους στόχους που μας απασχολούν εδώ. Στον τομέα της ελίας και πέραν αυτό, όταν είναι δυνατό να προσθέσουμε ότι ελευτικές ε, συμφωνίες με τις ε, τρίτες χώρες είναι μια εξαιρετική οδός για να θέσουμε σε εφαρμογή τους στόχους ε, της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής που φυσικά δεν μπορούν να περιοριστούν στον στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρμόζονται και πέραν των δικών μας συνόρων. Η δεύτερη σημαντική πτυχή έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Εδώ, η χρηματοδότηση των 50 μιλίων ευρώ που προτείνεται αναφέρεται παρά ε, το ότι ε, δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποσό. Δεν ε, φαίνεται επί του παρόντος ε, ότι είναι λογικό να ζητήσουμε ένα μεγαλύτερο κονδύλι. Έτσι λοιπόν αναφέρονται αυτά τα 50 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα είναι σημαντικό εδώ να ξέρουμε από πού προέρχεται το κονδύλι αυτό έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι δεν ε, θα αποσυρθεί επειδή θα έχουν χορηγηθεί άλλα κονδύλια στην Αλία. Η τρίτη πτυχή έχει να κάνει με την εγγύηση ε, της υιοθέτησης κατεξιοδότηση πράξεων. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν ε, πρέπει να χάσουμε. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικήσει τη κατεξουσιοδότηση πράξης, κάτι που έγινε και σε αυτή την πρόταση που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή. Και φυσικά αφού λάβαμε και γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας σε σχέση με το καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε να το πράξουμε αυτό και αφού επιβεβαίωσα ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Είμαι στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. En primer lugar, señor Antinori. Πρόεδρε, έφτασα με λίγη καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη. Έτσι δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στι ψηφοφορίε. Μήπως το μπορούσατε να καταγράψετε την παρουσία μου. Αν και στη μέσα διάταξη που είχα στη διάθεσή μου, οι ψηφοφορίε αναφέρονταν ότι θα διεξαχθούν στη νέα και το έρθω. Αυτά ήθελα να αναφέρω. Αργότερα θα ξαναλάβω το λόγο. Eh, Νομίζω πως η συνάδελφος ε, Πεδρανέβες έκανε μια εξαιρετική εργασία και ανέλησε την ουσία του θέματος ε, κάτι το οποίο συζητήθηκε στο παρελθόν όταν πρόκειτο να γίνει ε, κατανομή μέσα στην Επιτροπή και την ε, Επιτροπή Μεταφορών και πολύ καλά έκανε η Πρόεδρος που ζήτησε την ενισχυμένη συνεργασία. Συμφωνώ με τα όσα δήλωσε η συνάδελφος Νέβες εκτός από δύο-τρία θέματα και διαβάζοντας τις τροπολογίες ε, νομίζω ότι εδώ φάσκουμε και αντιφάσκουμε ή εγώ δεν καταλαβαίνω καλά ή τότε τα όσα άκουσαν τα αυτιά μου σήμερα αποκλίνουν. Αναφέρομαι σε μια λεπτομέρεια. Μιλάμε για ωκεανούς και ποτέ για θάλασσες ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε θάλασσες. Καταλαβαίνω πως απέναντι την Πορτογαλία υπάρχει ο ωκεανός, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη θάλασσα ή της Μεσογείου συγκεκριμένα. Θα μπορούσε να διορθωθεί λοιπόν αυτή η έλλειψη. Και έχω και δύο ενστάσεις επί της ουσίας ε, να πω ότι συμφωνώ με την αντιμετώπιση του θέματος, συμφωνώ ε, την αποκατάσταση της θέσης ε, της Αλίας στην πλαίσιο της ορκρομές θαλάσσιας πολιτικής αλλά εδώ δεν πρόκειται να ξαναγράψουμε τον κανονισμό για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, αλλά για την χρησιμοποίηση 50 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί δεν θέλαμε να, να διατυπώσουμε τον κανονισμό, τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε ευρύτερα το ζήτημα της θαλάσσιας πολιτικής και να είμαστε πολύ πιο κάθετοι στη σκέψη μα. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Μία αφορά στην τροπολογία υπαριθμών 16. όπου αναφέρονται προγράμματα και επεξήγησή τους, η οποία όμως δεν είναι ιδιαίτερα σαφής και δεν αφορά όλα σε όλα τα προγράμματα. Και δεύτερη παρατήρηση που είναι μάλλον ερώτηση. Στην έκθεση αναφέρεται πως είναι σημαντικές οι διεθνείς σχέσεις, αλλά στις τροπολογίες 18, 19 και 20 υπάρχει μια ουσιαστική κατάργηση των ζητημάτων που άπτονται των διεθνών σχέσεων. Κοιτάξτε, στη Μεσόγειο τώρα, σε όλη τη Μεσόγειο, δίχως ε, μια ολοκλήρωση και μια ενίσχυση των σχέσεων με τρίτες χώρες, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Υπάρχουν 7 κοινωνικέ χώρε ε, στην ε, Μεσόγειο και καμιά δεκαριά μη κοινωνικέ. Εξάλλου, η εδαφική συνέχεια έχει ως αποτέλεσμα πως αν δεν υπάρξει αυτή η ενίσχυση των ε, σχέσεων, τότε θα έχουμε αποτελέσματα τραγικά. Δεν αναφέρομαι τώρα σε ό,τι συμβαίνουν ανάμεσα στην Σικελία και τη μάλλον την Ισπανία και το Μαρόκο Αλγερία. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι ε, έχουμε αποστάσεις 30 ε, χιλιόμετρων, βλέπουμε τι συμβαίνει, διότι έχουμε δύο κοινέ χώρες, την Κροατία και την Ιταλία, η Σλοβενία και η Ιταλία που είναι κοινωνικέ χώρες και μία μη κοινωτική χώρα, η Κροατία, βρίσκονται στην ίδια λεκάνη που και που εισαπέχουν 50 χιλιόμετρα από την περιοχή. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε μια οπτική γωνία που θα συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς σχέσεις. Εξαιρετική εργασία της συναδέλφου. Δεν νομίζω ότι είναι πολλές οι τροπολογίες αν και η ίδια δήλωσε πως ε, είναι πολλές ε, και κάτι ακόμα το παράρτημα εμείς βρισκόμαστε ενώπιον των 50 εκατομμυρίων ευρώ που και η Κομισιόν προτείνει να, να τεθούν στο παράρτημα και στον κανονισμό. Αυτό είναι ένα θέμα κλειδί, διότι όταν εγκριθεί ο κανονισμός, οι γραμμές, τότε το παράρτημα ε, μπορεί μονόπλευρα να το τροποποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τα ποσά, τα κονδύλια να ε, δεσμευτούν περισσότερο με το κείμενο το οποίο θα εγκρίνουμε στην Ολομέλεια. Αναφέρω λοιπόν κάποιες τροπολογίες που θα αφορούν την μεταφορά κάποιου περιεχομένου του παρατήματος στο διατακτικό του κανονισμού. Εγώ συζήτησα με άλλες επιτροπές που συνεργάζονται, με τις οποίες συνεργάζονται ε, επ' αυτού του θέματος ε, και ενδεχόμενα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού θα βρούμε το περιεχόμενο αυτών των ε, λεγόμενών μου και κάτι ακόμα, να ζητήσω συγγνώμη από τις αλφωνεύες η γραμματεία κατάλαβε, δεν κατάλαβε καλά. Εγώ ζήτησα να προτάξουμε την έκθεσή σας, διότι πρέπει να πάω στην μεταφορών για να συζητήσουμε το ίδιο ζήτημα. Εγώ είμαι ο υπέτειος λοιπόν. Με συγχωρείτε, αλλά εμένα μου είπαν ότι η κυρία Πατράου είχε ζητήσει αυτήν την αλλαγή. Τέλο πάντων είναι ο κύριο Μιλάνα, δεν έχει σημασία. Ο κύριο Καντέκ. Oui, je reste, Madame la Présidente. Ευχαριστώ. Εγώ θα μείνω. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία και την εργασία της. Πολύ ενδιαφέρουσα για τις χώρες μας και για τις περιφερειές μας. Εγώ είμαι από τη Βρετάνη με πολύ έντονη θαλάσσια, όπως ξέρετε, ταυτότητα και η οποία βεβαίως ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ολοκληρωμένη πολιτική στον τομέα της αλίας. Αυτό μας αφορά όχι μόνο όσον αφορά τη θαλάσσια πολιτική, αλλά και όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής μας και τον σύνδεσμο που προσπαθούμε να πετύχουμε τον καλύτερο τρόπο μεταξύ των θαλάσσιων και των χερσαίων μεταφορών. Πολλοί συνάδελφοι έχουν στηρίξει την πολιτική για το Ατλαντικό τόξο. Όντως, ο Ατλαντικός είναι ωκεανός και όχι θάλασσα και εδώ είναι σωστή ορολογία. Αυτή η στρατηγική για τον Ατλαντικό θέλει κατά κάποιο τρόπο να συνδέσει την περιφερειακή πολιτική, περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Και βεβαίω η αλληλεία είναι εδώ μια πάρα πολύ σημαντική συνιστός αυτής της πολιτικής. Η συγγήτρια θα πρέπει να μην ξεχάσει αυτές τις πρόπτικες και αυτές τις προτεραιότητες που είναι διαφορετικές για την Μεσόγειο και για την περιοχή του Ατλαντικού. Θα πρέπει επίσης να προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί η θαλάσσια στην ιστόσα όχι μόνο αυτών των περιοχών αλλά όλης της Ευρώπης. Και εδώ θα ήθελα ιδιαίτερα να σκεφτώ τις offshore αναπτύξεις των πάρκων αιωλικής ενέργειας, κάτι που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες ακόμα περισσότερο δεδομένων των γεγονότων που συμβαίνουν εκτός Ευρώπης αυτές τις ημέρες. Πέρα λοιπόν από την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, την οικονομική ανάπτυξη, την αλία, τις ηχθειοκαλλιέργειες και στηρίζω ιδιαίτερα εδώ όλα τα πιλωτικά προγράμματα που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι αυτή η γνωμοδότηση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή Επιτσουσίας Είχαμε πολύ πρόσφατα μία εμπειρία μίας γνωμοδότησης, την οποία αγνόησαν παντελώς και το λέω πολύ ευγενικά. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο και με αυτήν την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ευχαριστήσω τη Μαρία για την πολύ καλή της έκθεση. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί μας ενημέρωσε ότι αυτή η γνωμοδότηση ενσωματώθηκε στην ενισχυμένη συνεργασία γιατί το 2006 όταν ξεκίνησε το θέμα αυτό η Επιτροπή Μεταφορών κατά κάποιο τρόπο πήρε τον ηγετικό ρόλο. Από ό,τι φαίνεται εδώ διαπιστώνεται η τρίτη θέση της αλίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως τα πλήγματα που γνωρίζουν οι αλληλείς μας καθημερινά είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Η Μαρία βεβαίως ε, μιλά για την ολοκληρωμένη πολιτική που είναι απαραίτητη λέγοντας ότι βεβαίως πρέπει να έχουμε μία λήψη αποφάσεων με συνοχή και σύμφωνα με τον κύριο Μιλάνο ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις παράκτιες περιοχές. So, I know from... Uh, Γνωρίζω, γιατί έχω την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου και την πίεση που έχουν υποστεί οι αλληλείς όσον αφορά την προστασία των παράκτιων περιοχών και πολύ συγκεκριμένων περιοχών με αποφάσεις που λαμβάνονται από πάνω προς τα κάτω και επιβάλλονται στους αλείς και πολλές φορές χωρίς καμία διαβούλευση με τους αλείς κάθε φορά που υπάρχουν θέματα ενέργειας, προστασίας ελλειμμάτων, προστασίας κάποιων περιοχών. Η επιθυμίες, αν θέλετε, αυτών των φορέων και αυτών των τομέων φαίνεται να επικαλύπτουν και να επιβάλλονται στους αλληλείς και αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να συντονίσουμε τις πολιτικές μας και βεβαίως να γίνει μια κοινή εκτίμηση όλων των συμφερόντων και των περιοχών αυτών και να μην προσπαθούμε απλώς να δημιουργήσουμε έναν πράσινο παράδεισο Υπάρχει επίσης και το 30% παραγωγής ε, ενέργειας αυτών των μονάδων καθ' όλη τη διάρκεια ζωή τους. Η αλήθεια είναι όμως ότι μόνο 20% αυτής της ενέργειας ε, παράγεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα δαπανώνται τεράστια ποσά, σπαταλώνται θα έλεγα μάλιστα τεράστια ποσά και την ίδια ώρα δεν μπορούν οι αλλοί να χρησιμοποιήσουν τεράστιες περιοχές, παραδείγματος χάρη ε, στο νότιο τμήμα της Σκοτίας, στην ε, νήσο Τάιρι, αποκλείεται μια περιοχή τεράστια, πιο μεγάλη από το ίδιο το νησί που είναι 6 χιλιόμετρα από τις ακτές. Όλη αυτή η περιοχή για γενιές αποτελούσε την περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν γενιές αλλιέων. Σήμερα αποκλείεται αυτή η περιοχή και το 2020 έχουν τεθεί ε, στόχοι για τις ε, νέες πηγές ενέργειας. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο πράσινος παράδεισος στον οποίο όλοι θέλουμε να φτάσουμε, αλλά ας κοιτάξουμε και την οικονομική συνιστόση αυτών των αποφάσεων. Όπως είπε και ο Αλακαντέ, Πρέπει να κοιτάξουμε την ανάπτυξη, πρέπει να κοιτάξουμε την ε, δυνατότητα δημιουργίας ε, νέων πηγών ενέργειας, τα κύματα παραδείγματο χάρη. Αλλά ας κοιτάξουμε και τις επιδοτήσεις, τα τεράστια ποσά που δίνονται, τριπλάσια ποσά που δίνονται, για να αναπτυχθούν αυτές οι νέες ε, πηγές ενέργειας. Η εναλλακτικέ, οι οποίε, επαναλαμβάνω, στοιχίζουν τρει φορέ παραπάνω από τι παραδοσιακέ αυτέ του άνθρακα. Οι αλλοί την ίδια ώρα παρεγκονίζονται και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η συγγήτρια έχει επισημάνει αυτό στην έκθεσή της. Και πραγματικά κάνετε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των αλλιών μας. Γιατί κάθε φορά βλέπουμε να αγνοούνται. Όλα αυτά τα χαιρετίζω ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Κύριε Βέμερς. Yeah, Ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για τις αλλαγές αυτής της έκθεσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης που βλέπω ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν λόγο. Θα πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί σε αυτές τις προτάσεις. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι σήμερα θα πρέπει να εξετάσουμε και τις περιοχές της επιφάνειας της θάλασσας έτσι όπως έχουν καθοριστεί. Δεν πρέπει να είμαστε άκαμπτοι. Ε, οι αλίες καταλαβαίνετε ότι δεν τοποθετούνται κάπου στη θάλασσα και δεν κουνάνε από εκεί σαν τις αγελάδες σε ένα χωράφι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ευελιξία στον καθορισμό των περιοχών. Επίσης, η χρηματοδότηση. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης. Σε ποιες πολιτικές απευθύνονται. Τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο έχουν αποφασιστεί. Επίσης, να δείξουμε σύγχρονο πνεύμα. Όντως υπάρχει η πράσινη ε, τάση η παραδοσιακή και νέα χρησιμοποίηση των ε, θαλάσσιων πόρων. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης ε, να συνεχίσει να έχει τα δικαιώματά του όσον αφορά τη συναπόφαση, καθώς και τις ε, κατοικιοδότηση πράξεις, θέμα που συζητήσαμε. Πραγματικά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι οι θάλασσες, οι θαλάσσιες περιοχές να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αυτής της ολοκληρωμένης πολιτικής για τις θάλασσες και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν όλοι βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι. Κύριε Λεβίν. Κυρία Λεβίν, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της. Για τα σχόλια του κυρίου Στίβενσον. Νομίζω ότι πίσω από την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική εναπόκειται η ιδέα ότι προσπαθούμε να λάβουμε κάποιες λογικές αποφάσεις για το πώς να χρησιμοποιήσουμε πιο υφόρο τρόπο το βυθό της θάλασσας έτσι ώστε να υποφεληθεί όλη η κοινωνία στο σύνολό τη. Νομίζω ότι αυτή είναι η ιδέα που αναπόκειται πίσω από αυτό, αλλά ακριβώ αυτό θέλω να ρωτήσω και την κυρία Πατρόνεδε. Εξέτασα την τροπολογία 7 και την τροπολογία 7 της Επιτροπής Μεταφορών, όπου λέγεται ότι ο στόχος της ολοκληρωμένης, θα, αναφέρει το στόχο της ολοκληρωμένης πολιτικής, αλλά έχει διαφορετικό ορισμό η κυρία Πατρονέβες από τον ορισμό που χρησιμοποιεί η Επιτροπή Μεταφορών. Να το διαβάσω. Λέει ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο ξεσκαλούμενο το πρόγραμμα Πρωτορχικό στόχο του οποίου είναι η μεγιστοποίηση της βιώσιμης εκμετάλλευση των πιο απομακρυσμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συσχετιζόμενων πολιτικών και της ε, διεθνούς σχετικής συνεργασίας. Διάβασα την τροπολογία της Επιτροπής Μεταφορών, ενώ η κυρία Πετρολέμης λέει πρωταρχικό στόχος ε, είναι η μεγιστοποίηση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλασσών και των ωκεανών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας και των παράκτων περιοχών. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, δηλώνεται πουθενά ποιος είναι ο στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι ο ορισμός, όπως έχει διατυπωθεί από την κυρία Πατράων ουσιαστικά μα δεσμεύει υπερβολικά. Δηλαδή, όταν λέμε χωρί να τη κίνδυνο ανάπτυξη θελέσσια οικονομία και των παράκτων περιοχών, Δηλαδή, ποιο ακριβώ είναι ο στόχο τη ολοκληρωμένη θελέσσια πολιτική, κυρία Πατράου, να δείτε πώ μπορείτε να μα το εξηγήσετε αυτό. Και επίση το θέμα των 50 εκατομμύριων ευρώ. Ξέρει η συγγήτρια από πού προέρχεται αυτό το κονδύλι. Είναι μια γενική ερώτηση. Έχετε μια απάντηση σχετικά με αυτό που προέρχεται το κονδύλι. Κύριος Γκροβερτσίκ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να δηλώσω πως υποστηρίζω την ε, έκθεση και Συμφωνώ με τις εργασίες ε, της συναδέλφου Πατράου Νέβες, ε, διότι όπως ε, ακούσαμε η έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και για το Ευρωκοινοβούλιο σύνολό του, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχει απουσία αυτής της ολοκληρωμένη θαλάσσιας πολιτικής και αυτή είναι μια απουσία, μια έλλειψη που γίνεται αισθητή σε όλα τα κράτη-μέλη έχει επιπτώσεις ε, στην οικονομία των παράκτιων περιοχών. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στα όσα ανέφερε η κυρία Πατράου Νέβες. Η έκθεση της τροποποιείται ε, αισθητά μέσω των τροπολογιών. Αλλάζει η ίδια η δομή της έκθεσης. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε μια κοινή θέση, μια θέση στεναρή, την οποία θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε στο πλαίσιο της Επιτροπής Μεταφορών. Διότι δεν θεωρώ πως η Επιτροπή Μεταφορών εύκολα θα υποχωρήσει και θα δεχθεί όλες τις τροπολογίες και δεν φαντάζομαι ότι ιδιαίτερα θα δεχθεί τις τροπολογίες της δικής μας Επιτροπής που ετέθη σε δεύτερη μοίρα και δεν έχει ακουστεί η φωνή μας μέχρι τούδε αυτό λοιπόν δηλώνω ότι στηρίζω την εισηγήτρια, αλλά να υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντική η κοινή μας θέση επί της εκθέσεως αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μια διευκρίνηση και μια παρατήρηση για τα 50 εκατομμύρια. Εγώ είμαι σκιώδης στους προϋπολογισμούς για αυτή την έκθεση. Αυτό ουσιαστικά προέρχεται από το κεφάλαιο 2, δηλαδή η γαλλωτική ανάπτυξη και η γεωργία. Αυτά τα 50 εκατομμύρια θέλουμε να ενσωματωθούν όχι στο παράρτημα του εγγράφου, αλλά στον κανονισμό, έτσι ώστε να ενισχυθεί. Το δεύτερο σημείο είναι ότι υποβάλλουμε μια τροπολογία που πιστεύω θα στηριχθεί Όσον αφορά τη νομική βάση αυτής της ε, θαλάσσια ολοκληρωμένης πολιτικής, μετά το 2013, γιατί όλοι ξέρουν ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα θα τεθεί κυρίως μετά το 2013. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν για τα αιωλικά πάρκα, τα offshore αιωλικά πάρκα, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική έχει σαν σκοπό να υπάρξει συνεργασία και όχι αντιπαράθεση μεταξύ δραστηριοτήτων. Είναι πιο δύσκολο βεβαίως να βρούμε συνεργασία και παράγοντες συνδυασμού παρά την αντιπαράθεση. Εγώ προέρχομαι από ένα τομέα όπου οι αλείς μπόρεσαν να δεχτούν αυτά τα αιωλικά πάρκα offshore κατάφεραν να δουν, αν θέλετε, τα οικονομικά συμφέροντα που απορρέουν για αυτούς από αυτά τα ε, παράκτια πάρκα. Ας μην είμαστε λοιπόν πάντα απόλυτοι. Υπάρχουν συνδυασμένα συμφέροντα πολλές φορές και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των αλλιέων και των offshore αιωλικών πάρκων, κάτι που είναι για μένα πολύ απλοϊκό. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγητρία για την εκπόνηση της έκθεσης για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ε, και φυσικά δεν είναι κάτι πρόωρο γιατί θα πρέπει ε, να σκεφτούμε εκ των προτέρων δεν μπορούμε να έχουμε κατακαιρματισμένες πολιτικές γιατί φυσικά ξέρετε ότι δεν υπάρχουν γεωγραφικά ή πολιτικά σύνορα στους ωκεανούς έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε μια τέτοια πολιτική και καλό είναι να τη θέσουμε τον νωρίτερο σε εφαρμογή. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρξε η διευκρινήση για τα 50 εκατομμύρια, γιατί είχα και εγώ αυτή την ερώτηση. Ήταν πολύ ασαφέ από πού προέρχονταν διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε οποιοδήποτε νούμερο και να ελπίζουμε να έλθει από, το αποθεματικό. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί και τμήμα του κανονισμού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική και σκέφτομαι κυρίως τα πλεονεκτήματα. Φυσικά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα ε, της ανανεώσιμης πηγές ενέργειας ε, λόγου χάρη υπόθηκε το ότι ίσως ε, από τα offshore θα πρέπει να έλθει το 80% μέχρι το 2020 στον τομέα της ενέργειας. Όμως είναι σημαντικό και για την ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουμε μια στρατηγική γιατί έχουμε αλληλείς που εξαρτώνται πάρα πολύ ε, από την αλληλία, αλλά μπορούν όλοι αυτοί να εργαστούν δίπλα-δίπλα και τελικά να ωφεληθούν όλοι. Έτσι λοιπόν και η διαβούλευση είναι σημαντική και η κοινή λήψη αποφάσεων είναι σημαντική και συμπερίληψη των 50 εκατομμυρίων θα πρέπει να υπάρχει στο διατακτικό και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ. Ένα σχολείο πολύ γενικό. Πολλοί προλαλήσαντες είπαν ότι αυτή η στρατηγική έχει κάποιους κατάλληλους στόχους, ε, σημαντικούς, ευρύς. Θα έλεγα ότι το ποσό που προτείνεται για την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής, δηλαδή τα 50 εκατομμύρια, θα ε, μπορούσε να απορροφηθεί το ποσό αυτό από οποιαδήποτε γραμμή δάση που προτείνεται. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση για το ποσό που διατίθεται για την στρατηγική αυτή. Εμείς πάντοτε είχαμε ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της στρατηγικής. Ε, λέγαμε πάντοτε ότι σε νέους στόχους πρέπει να ανταποκρίνεται και νέα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Τώρα, αυτό που προτείνεται εδώ είναι για ένα προσωρινό μέχρι το 2013 και έχουμε ένα κονδύλι 50 εκατομμυρίων που θα χρησιμοποιηθεί σε μία βάση συγχρηματοδότησης, δηλαδή και τα κρατημέλη πρέπει να συμμετέχουν. Αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω εγώ. Ότι αν και αυτή είναι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, θα πρέπει εδώ να ε, είμαστε προοριοσμένοι, γιατί αυτός ο ορίζοντας ε, απαιτεί την ίδια χρηματοδότηση ε, κοιτάξτε, βλέπουμε τι περιορισμοί έχουν ε, ε, ληφθεί, τι περικοπές έχουν γίνει σε διάφορα κράτη, όπως στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, κράτη που θα ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για την ανάπτυξη αυτή της στρατηγικής και ουσιαστικά βιώνουν κάποια καθεστώτα λιτότητας και μειώνονται υπερβολικά τα δημοσιοοικονομικά. Έτσι λοιπόν μπορούσα να μιλήσω εδώ για όλα τα υπόλοιπα που προβλέπετε σε αυτά τα σχέδια και στην Πορτογαλία ανακοινώθηκαν ε, νέα μέτρα αυτή τη βδομάδα στην Πορτογαλία. Εγώ νομίζω ότι ε, τα κράτη που εποφελούνται από την εσωτερική αγορά ε, μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν αυτά κονδύλια όμως εδώ τελικά αντιτιθόμαστε σε, αντιτιθέμεθα σε αυτούς τους στόχους όταν ε, ε, λέμε ότι ε, εδώ τελικά πρέπει να προωθήσουμε την οικονομική συνοχή. Πώς θα το κάνουμε αυτό, γιατί ε, όσοι χρειάζονται περισσότερο αυτή τη στρατηγική τελικά είναι αυτοί που θα υποφεληθούν λιγότερο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των στόχων αυτής της πολιτικής και της νέας χρηματοδότησης που προβλέπεται και της πραγματικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που πάρα πολύ συγκεκριμένα είπε ο κύριος Κάλικα όσον αφορά την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Μιλάμε για τις μεταφορές και μιλάμε για τους αλείς, για την αλία, ενώ δεν υπάρχουν καθορισμένες αρμοδιότητες. Σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών, εξάλλου πρέπει να πάω, υπάρχει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Εμείς, σαν Επιτροπή Αλίας, πρέπει να θέσουμε με σαφήνεια ποια είναι τα σημεία και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Τα σημεία αυτά, τα οποία σαφώς πρέπει να διατυπώσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όταν μιλάμε για αλία, όταν μιλάμε για αλλιευτικά σκάφη, για κυκλοφορία αυτών των σκαφών. Βεβαίως υπάρχουν θέματα μεταφορών, θαλάσσιων μεταφορών, αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε και την οργάνωση αυτών των θαλάσσιων περιοχών και πώς θέλουμε στο μέλλον να γίνει η χρησιμοποίηση αυτών των πόρων. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, Υπάρχει το θέμα της ενέργειας, ε, υπάρχουν οι τροφοδοσίες, ε, οι προβλέψεις για τις μεταφορές και όντως υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των διαφορετικών τομέων της χρήσης των ε, πόρων και όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις που γνωρίσαμε τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές. Η στρατηγική λοιπόν και ο καθορισμός της είναι ο δικός μας τομέας και πρέπει σαφώς να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε και να επιμείνουμε στα σημεία αυτά που θέλουμε να προωθήσουμε σαν Επιτροπή Αλληλείας και σαν τροπολογίες και πολλές φορές υπάρχουν ε, διαφορετικά συμφέροντα. Πολλές φορές το θέμα της ασφάλειας των λιμένων που αφορά και την Επιτροπή Μεταφορών αλλά και τη δική μας μπορεί να είναι εξάλλου κοινά σημεία. Μα δεν θέλει κανείς ε, να μπλεχθεί στα πόδια άλλων ε, σε ό,τι αρμοδιότητες. Εδώ εφαρμόζουμε το άρθρο 50 και σε αυτό το πρόγραμμα όπου ήταν πολύ δύσκολο να διαχωρίσουν ποια είναι τα αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών και της Επιτροπής Αλίας, τελικά αποφασίστηκε και οι δύο επιτροπές θα έπρεπε να εξετάσουν το ζήτημα, αλλά βρισκόμαστε σε μια αρχική ακόμα Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ξεκάθαρη και λοιπόν όλοι οι τομείς που έχουν σχέση με την ε, θάλασσα εμπλέκονται και στο Καροκάρι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, επί τη εκθέσεω ε, Πατράου μεταξύ ημών και τη Επιτροπή Μεταφορών. Να κάνω κάποια σχόλια τώρα και μια σειρά από ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σε αυτή τη φάση ε, είμαστε στην αρχική φάση, τα προπαρασκευαστικά ολοκληρώθηκαν, αλλά αυτή είναι η δεύτερη φάση και θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. αυτό το ζήτημα το δημοσιονομικό. Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν δαπανήθηκαν τα κονδύλια που βλεπόνταν στην προπαρασκευαστική φάση, διότι θεωρώ ότι η χρήση των κονδυλίων δεν ε, εξαντλήθηκε. Και τώρα σε ό,τι φορά τα 50 εκατομμύρια που προβλέπονται για αυτό το νέο πρόγραμμα, όπως το ονομάζει η Κομισιόν, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ζήτημα του περιθωρίου που δεν είναι ξεκάθαρο. Στην πρόταση της Επιτροπής το δημοσιονομικό δελτίο δεν είναι ξεκάθαρο και αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο που αναλογεί στην αλία και τι θαλάσσιες υποθέσεις ε, που προέρχεται το κεφάλαιο 11, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το ζήτημα έτσι ώστε στο μέλλον να μην οδηγηθούμε σε μείωση των κονδυλίων τώρα. Κάτι ακόμα. Έχω μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό ρωτάω την Κομισιόν σχετικά με το ζήτημα της επιτροπολογίας. Έχω τις εμβολίες μου που οι κατεξόδοτες πράξη είναι καταλληλότερες σε αυτήν την φάση. Τροπή Μεταφορών αλλά και η έκθεση Πατράου ε, ε, ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 290 και όχι συμβουλευτική επιτροπή όπως προτείνει η Κομισιόν, αλλά νομίζω ότι η πρόταση των κατεξιόδων πράξεων είναι μάλλον υπερβολική. Θα ήθελα λοιπόν, ε, γιατί η κυρία Πατράου δέχθηκε το θέμα αυτό. Κύριε Πατράου, έχει το λόγο. Ε, Συγγνώμη, κυρία Μπενίνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα όλα τα μέλη της Επιτροπής για το ενδιαφέρον που δείχνουν για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Πιστεύουμε ότι η πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν υπάρξει πλήρη στήριξη αυτών των στόχων για μια πιο συνεκτική χρήση ε, των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων. Πιστεύουμε ότι όλες οι δραστηριότητες ε, στη θάλασσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με έναν ε, βιώσιμο τρόπο και ιδιαίτερα κάποια από τα σημεία που αναφερθήκατε εδώ όπως παραδείγματο χάρη πώς υπάρχει ένα σχετικός ανταγωνισμός μεταξύ όλων αυτών που ζουν και χρησιμοποιούν την θάλασσα. Προτείνουμε λοιπόν εδώ έναν μηχανισμό σχεδιασμού των θαλασσών και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι στον σχεδιασμό αυτό όλες αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζονται με διαφάνεια, λαμβάνοντα υπόψη όλες τις απόψεις, όλες τις θέσεις και όλα τα συμφέροντα όλων των κοινοτήτων, όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις θαλάσσιες περιοχές, θα πρέπει να αναπτύσσονται με στόχους μακροχρόνιους και βιώσιμους. Με αυτόν τον τρόπο και αν στοχεύσουμε στην ανάπτυξη και στη συνέχεια αυτής της πολιτικής, πιστεύω θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Πώς δαπανώνται τα χρήματα, αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που ακούστηκαν. Τα χρήματα δαπανήθηκαν, και αυτό είναι πολύ θετικό, για τους στόχους και τις πολιτικές για τις οποίες είχαν δεσμευτεί και αυτό συνεχίζεται για τα ποσά που βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία. Τα ποσά που έχουν χορηγηθεί σε εμά για την προετοιμασία και τα πιλωτικά προγράμματα έχουν δαπανηθεί για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν δει. 20.461.933 για το 2008-2010 οι λεπτομέρειες των δαπανών θα παρουσιαστούν, θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όλες οι λεπτομέρειες για τα πιλωτικά προγράμματα και την προετοιμασία θα χορηγηθούν. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας, γιατί προτείνεται μια συμβουλευτική επιτροπή, θα απαντήσω ότι ο κανονισμός θέτει καταρχήν την προετοιμασία του πώς θα δαπανηθούν τα συγκεκριμένα ποσά μέσω των πιλωτικών προγράμμων κατόπιν, οι συγκεκριμένες δράσεις για το 2010, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, και σύμφωνα με τα στοιχεία και τη γνώση που διαθέταμε τότε μεταξύ του 2010 και σήμερα, αλλά και αύριο, από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί και θα προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως έχουμε ολοκληρώσει την προετοιμασία, τα πιλωτικά προγράμματα και έχουμε νέες πληροφορίες και μεγαλύτερη γνώση. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτά τα μαθήματα, σε αυτά τα οποία μπορέσαμε να μάθουμε από την προετοιμασία, από τα πιλωτικά προγράμματα και να εμπλουτίσουμε και να ενημερώσουμε και να βασίσουμε την παρούσα δράση μας σε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν μια συμβουλευτική επιτροπή. Πρώτον, γιατί πρόκειται για κάτι που δεν στοιχίζει ε, πολύ. Αν θυμάστε, βάσει της επιτροπολογίας, σήμερα δεν έχουμε ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα. Άρα, ε, το σημαντικό ποσό που θα χρειαζόταν για μια κανονιστική επιτροπή δεν υφίσταται, γι' αυτό και ζητάμε την συμβουλευτική. Και επιπλέον πρόκειται για την υλοποίηση ενός ετήσιου προγράμματος εργασιών για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε την βασική πράξη ή να υλοποιήσουμε ε, τους στόχους έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε. Η κυρία Πατράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους στοχους ετσι οπως εχουν παρουσιαστει και αυτο πιστευω οτι πρεπει να κανουμε η κυρια Πατρά. ευχαριστω προεδρε ευχαριστω και ολους τους συναδελφους για τα σχόλιά τους ε, και για ορισμένες από τις ερωτήσεις που μου έθεσαν, καθώς μου δίνουν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ορισμένα σημεία που σε μεγάλο βαθμό ήδη αναφέρονται στην ίδια την έκθεση. Καταρχήν να υπογραμμίσω κάτι που αναφέρθηκε εδώ, ότι στο θέμα που μας απασχολεί σήμερα εμείς ε, μόλις μιλάμε για τη χρηματοδότηση και όχι για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αυτή καθ' αυτή διαφορετικά θα είχαμε πολύ περισσότερα να πούμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε σε ποιο πλαίσιο βρισκόμαστε και πράγματι από τώρα, από το τέλος του 2010 μέχρι το 2013 αναφερόμαστε στην ε, χρηματοδότηση και γι' αυτό μιλάμε για τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ορισμένοι συνάδελφοι ρώτησαν ε, από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά. Αναφέρεται με πολύ μεγάλη σαφήνεια στην τροποποίηση 32. Έτσι λοιπόν σας παραπέτω Εκεί λέει συγκεκριμένα βάσει του περιθωρίου που αναφέρεται στον τομέα 2. Αυτή είναι η προέλευση λοιπόν της χρηματοδότησης. Δεν υπάρχουν ε, μεγάλες αμφιβολίες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ε, βάσει όλων των πληροφοριών που είχα εγώ για το από πού προέρχονται τα χρήματα για τα οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή. Και επίσης ποιος είναι ο προορισμός. Προορίζονται για μια σειρά δράσεων που ανακοινώνονται με έναν οργανωμένο τρόπο από την τροπολογία 25. Από εκεί και πέρα έχουμε μία σειρά τομέων όπου θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Πιστεύω ότι η διατύπωση είναι αρκετά ευρεία έτσι ώστε ε, να καλύψει τις προτάσεις που ακούστηκαν. Σε αυτή τη διατύπωση προσπαθήσαμε το εξής, ε, να είμαστε αρκετά συγκεκριμένοι για το πού θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα, σε ποια είδη δράσεων, αλλά δεν θέλαμε να είμαστε και περιβολικά περιοριστικοί έτσι ώστε να μπορούμε να συμπεριλάβουμε και διάφορα άλλα project που θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτά τα 50 εκατομμύρια. Νομίζω ότι κυρίως αυτές οι ερωτήσεις τέθηκαν σχετικά με τη χρηματοδότηση. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έθιξαν διάφορες συνάδελφοι είχε να κάνει με το να προχωρήσουμε με σαφή τρόπο για ολοκληρωμένες, δεδομένε πολιτικές και να μην ε, υπάρχει κατακαιρματισμένη πολιτική. Να απορρίψουμε την κατακαιρματισμένη πολιτική. Φυσικά δεν μιλάμε για ολοκληρωμένη θαλασσία πολιτική, ακριβώς αυτό είναι ο στόχος. Αφενός να έχουμε ένα ευρύ όραμα ε, για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, να γνωρίζουμε όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκεί και με ένα διαρθρωμένο τρόπο να επιτρέψουμε οι δραστηριότητες αυτές πράγματι να καταλαμβάνουν τον απαραίτητο χώρο. Θα ήταν εξαιρετικό αν ήδη μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε την επικρατεία της θάλασσας. Ο στόχος όμως ε, είναι να είναι διαρθρωμένες όλες αυτές οι δραστηριότητες και με έναν άτυπο τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα σύστημα από πάνω προς τα κάτω, αλλά να υπάρχει μια συμμετοχή όλων όσων έχουν συμφέροντα στη θάλασσα έτσι ώστε να μπορούν να διαρθρωθούν αυτές οι πολιτικές. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εξαρτάται και από την οργάνωση των ίδιων των κρατών μελών και από οργανισμούς που δημιουργούνται, που συσταθεί για να λάβει η χώρα αυτή η επίδραση. Γιατί εδώ έχουμε μεικτές αρμοδιότητες. Αλλά να επανέλθω στο ουσιαστικό θέμα εδώ, που είναι ότι θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν χώρα όλες τις δραστηριότητες, ε, δίχως ε, να ζημιώνεται η μία ή η άλλη. Και επίσης θα πρέπει να τις ξανασχεδιάσουμε. Να λάβουμε υπόψη και τους προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πέρα αυτού και να λάβουμε υπόψη τι πολιτική χαράσουν οι οργανισμοί που συστήνουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά αυτή η πολιτική. Όταν ε, μιλάμε για τις διορθωμένες πολιτικές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμπλέκοντας και διάφορες επιτροπές ε, και είναι και με δικός μας στόχος Τη ε, δική μας επιτροπής, να έχουμε το καθεστώ τη συνδεδεμένη επιτροπή. Τι νόημα θα έχει μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που δίνει ένα προσδελισμό για την κοινή χρήση των ωκεανών και των θαλασσών και να είναι μόνο μια επιτροπή αρμόδια για όλο αυτό το θέμα. Έτσι θα προδίδαμε όλο το πνεύμα τη ολοκληρωμένη θαλασσίας πολιτικής. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών Ελίας και Μεταφορών για να πετύχουμε ακριβώς μια καλύτερη διάρθρωση για την χρήση των θαλασσών. Για το θέμα αυτό πιστεύω ότι με την Επιτροπή Μεταφορών θα είναι δυνατόν να φτάσουμε σε ευρεία συνένεση. Μάλιστα, μια συνεδρίαση όλων των ε, ενεχομένων επιτροπών ε, στην έκθεση αυτή ε, κυριάρχησαν οι συμβιβασμοί, ε, συνομιλήσαμε και με τον αρμόδιο εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών και όλα μου οδηγούν στο να πω ότι θα είναι δυνατό να έχουμε εδώ ένα κοινό προσανατολισμό. Τώρα, σας υπόθηκαν για την τροπολογία 7 ότι είναι αντιφατικέ οι δύο τροπολογίε τη δική Επιτροπή και τη Επιτροπή Μεταφορών. Δεν το δέχομαι ότι είναι αντιφατικέ. Ε, πιστεύω ότι είναι διαφορετικέ, ναι. Όμω ε, ξεκινάμε από διαφορετικά σημεία εστίαση. Ε, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Πιστεύω όμω ότι όταν συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Μεταφορών θα μπορέσουμε συμπληρωματικά να φτάσουμε σε μια κοινή πρόταση. Αυτή τη στιγμή δεν αναμένω να υπάρξουν μεγάλες δυσκολίες. Μία τρίτη πτυχή που αναφέρθηκε επίση από δύο φορές συναδέλφου, έχει να κάνει με την αναγκαιότητα να συμμετάσχουν και άλλε χώρε πέραν τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πτυχή αναφέρεται στην έκθεση, συγκεκριμένα στι τροπολογίε 11 και 23, δηλαδή Αναφερόμαστε εκεί στην εξωτερική διάσταση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και φυσικά είναι προφανές για μας ότι οποιαδήποτε ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική πρέπει να εμπλέκει και άλλες χώρες πέραν των κρατών μελών, γιατί διαφορετικά θα καταδικαζόταν σε αποτυχία. Στην πρώτη μου παρέμβαση ανέφερα ότι η ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει να αποτελούν ένα διαβλό, μια ευκαιρία για να συμπεριληφθούν σε αυτές τις συμφωνίες το μέτρο του δυνατού το πνεύμα μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Πέραν αυτών των τριών πτυχών, που αναφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Υπήρξαν κάποιες λεπτομέρειες, ε, κάποια συγκεκριμένα θέματα σε ό,τι αφορά ότι γίνεται αναφορά σε ωκεανούς ελόχης της θάλασσης, ε, οι θαλάσσιες δραστηριότητες, ε, υπάρχουν στροπολογίες 2, 7, 10, 21... Δεν νομίζω ότι έχω παραλείψει την αναφορά στις θάλασσες. Βέβαια, επιφυλάσσομαι να ξαναδιαβάσω το κείμενο υπό το φως όλων των σχολείων που έγιναν εδώ. Σε κάθε περίπτωση, στην τροπολογία 16, Ακούστηκε το ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε ορισμένα project γιατί θα υπάρξουν και άλλα. Ναι, κοιτάξτε, αναμφισβήτητα. Στη τροπολογία δεξι αναφερόμαστε σε ορισμένα παραδείγματα. Και ίσως παραλείπονται κάποια άλλα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσθεθούν. Δεν έχω αμφιβολία. Έγινε και αναφορά στο τοπολογίες 18 και 20, όπου διαγράφονται σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Αναγνωρίζω ότι αυτή η πτυχή μπορεί να μην είναι αμέσω σαφή, αλλά αποτελεί με αυτού που είπα στην αρχή. Δηλαδή έχουμε καλύτερη οργάνωση του κειμένου εδώ. Ό,τι διαγράφεται εδώ βρίσκεται στις τροπολογίες ε, από την 23 και έπειτα. Δηλαδή δεν διαγράφουμε τίποτα ότι έχει να κάνει, σχέση με τι, ότι έχει να κάνει με τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Βάσει των σημείωσεων που έλαβα, πιστεύω ότι απάντησα σε όλα όσα μου παρουσιάσατε, εκτός από τις καταξουσιοδότηση πράξεις. Δεν αναφέρθηκε ακόμη σε αυτό. Εδώ, για δύο λόγους έγινε αυτή η επιλογή. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, ε, αρχή ε, που εκδίδουν προπολογισμό θα πρέπει να έχει λόγο σε ό,τι αφορά την ετήσια προεκοδότηση και το σχεδιασμό και εκτέλεση του χρηματοδοτικού κονδυλίου. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό μόνο στην Κομισιόν. Από την άλλη, ε, από τις συνεδριάσεις που είχαμε με τις υπόλοιπες ε, επιτροπές ε, προέκυψε ως κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε αυτό. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα, θυμήθηκα και κάτι που ξέχασα στο ότι ορισμένες συγκεκριτικές πτυχές υπάρχουν στο παράρτημα Αναφερθήκατε στην προέλευση της χρηματοδότησης. Στην ε, πρότασή μου εδώ δεν υπάρχει στο παράρτημα, αλλά στο διατακτικό του κανονισμού. Νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλια και επαναλαμβάνω ότι θα ξαναδιαβάσω το κείμενο υπό το φως των σχολείων και αν διαπιστώσω ότι υπάρχει κάτι που δεν έχει συμπεριληφθεί και χρειάζεται να συμπεριληφθεί θα το πράξω ευχαρίστω. Ευχαριστώ. A ver. Bueno, eh, quiero decirles και... Να σας πω πως... Ε, επειδή καταρτίζουμε αυτή τη γνωμοδότηση για τη διαδικασία του άρθρου 50, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Μεταφορών. Δεδομένη σημασία του θέματος, οι πολιτικές ομάδες ε, διαβουλεύθηκαν και συμφώνησαν πως η ημερομηνία για την τροπολογιών ε, κλείνει αύριο διότι υποχρεωτικά πρέπει να ψηφίσουμε την ελόγου δότηση στις 4 Απριλίου στο Στρασβούργο σε μια έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών Διαφορετικά δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα ούτε η δρομοδότηση ούτε οι τροπολογίε μα. Μισό λεπτό κύριε Αρσένη να εξηγήσω μερικά πράγματα. Καταλαβαίνω πως ε, αυτό δημιουργεί κάποια προβληματάκια για τους ε, βουλευτές αλλά και για μένα. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εάν ε, ορίσουμε διαφορετική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών θα μπορέσουμε να υποβάλουμε έγκαιρα την γνωμοδότησή μας, άρα όλος ο αγώνας που κάναμε για το άρθρο 50 πάει τζάμπα. Σας ε, παρακαλώ λοιπόν ε, να αξιολογήσετε το θέμα και νομίζω ότι αύριο το μεσημέρι πρέπει να είναι η καταληκτική ημερομηνία της τροπολογίου. Διαφορετικά τονίζω για μια ακόμα φορά ότι αγωνιστήκαμε για τίποτα. δεν θα χρησιμεύσει τίποτα. Πραγματικά θα κάνουμε την Επιτροπή Μεταφορών να μη διάσει. Κύριε Ασένη. First of Θα ήθελα να συγχαρώ την γραμματεία. Say in this very, very important... Είναι πολύ σημαντικό που και εμείς μπορούμε να εκφραστούμε σε αυτήν την προσπάθεια για νομοθεσία και για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Και εγώ είμαι εισηγητής μιας έκθεσης για το άρθρο 50 και σύμφωνα με το άρθρο 50. Εάν, εάν η γνωμοδότηση αυτή δεν ενσωματωθεί στην ψηφοφορία της Επιτροπής Μεταφορών, μπορεί να υποβληθεί εκ νέου στην Ολομέλεια βάσει του άρθρου 50. Ίσως λοιπόν, καλό θα ήταν να περιμένουμε να προετοιμάσουμε σωστά τις τροπολογίες, γιατί εάν για κάποιο λόγο δεν λάβουν υπόψη τους τις αποφάσεις μας, μπορούμε εκ νέου να τις υποβάλουμε στην Ολομέρα. Και με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσουμε την τελική μορφή της έκθεσης. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να πούμε στην Επιτροπή Μεταφορών να αναβάλουν την ψηφοφορία τους για να μπορέσουμε να εργαστούμε σωστά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτά, τα, σε αυτά τα οποία λέτε. Λοιπόν, εάν εμείς διατηρήσουμε αυτή τη δυνατότητα υποβολή στην Ολομέλεια, τότε ε, χάνουμε την δυνατότητα, εάν υπάρξει πρόβλημα με την υιοθέτηση τροπολογιών μας από την Επιτροπή Μεταφορών, τότε δεν θα έχουμε την εναλλακτική, της, ε, την εναλλακτική λύση που εσείς λέτε, δηλαδή να καταθέσουμε την Ολομέλεια. Διότι ξέρετε πολύ καλά πως μερικές φορές ε, υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την αποδοχή τροπολογιών μας από άλλες κοινοβουλευτικές τροπές. Λοιπόν, Εάν τυχόν προκύψει κάποιο πρόβλημα στην Επιτροπή Μεταφορών, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο λέτε εσείς. Και οι πολιτικές ομάδες ε, προτιμούν ε, να, τη λύση που εγώ προανέφερα. Εντάξει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά ε, το προτιμότερο είναι η δική μου πρόταση με τη δυνατότητα προσβήσει την Ολομέλεια όπως είπατε και εσείς σε ύστερο στάδιο. Εγώ θέλω να πω το εξής, εάν όλοι οι βουλευτές είναι αντίθετοι με αυτά τα οποία έχουν πει οι πολιτικές ομάδες, τότε μας το πούμε και θα συνεκολουθήσουν μια διαφορετική οδό. Κυρία Μπιλμπάου. συγγνώμη κυρία Ντεσμπαρέα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι διευκνήσατε κάπω τα πράγματα, αλλά να θέσω μια ερώτηση προ τη Γραμματεία. Εάν δεν υποβληθούν τροπολογίε μέχρι αύριο, μπορούμε να υποβάλουμε νέε τροπολογίε στην Ολομέλεια. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή όχι. Και αν δεν καταθέσουμε λοιπόν τροπολογίε αύριο, μέχρι αύριο μάλλον δεν θα έχουμε δυνατότητα να καταθέσουμε τροπολογίε στην Ολομέλεια. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Στην Ολομέλεια πάντα μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίε. Αλλά το πρόβλημα είναι πω ε, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 50, μόνο αυτέ ε, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αλίας ε, μπορούν να κατατεθούν στην Ολομέλεια, αλλά όχι με βάση το άρθρο 50. Λοιπόν, το άρθρο 50 αναφέρει ότι οι τροπολογίες πρέπει να έχουν εγκριθεί προηγούμενα. Αλλά εσείς σε προσωπικά μπορείτε να καταθέσετε ή οποιοδήποτε άλλο βουλευτή μπορεί να καταθέσει τροπολογίες απευθεία στην Κυρία Μπιλμπά, ευχαριστώ. Να ζητούσα την γνώμη των πολιτικών ομάδων. Να σας πω όμως ότι συμφωνώ με όσα είπατε. Εγώ είμαι μέλο τη Επιτροπή Μεταφορών και ζήτησα να ακολουθεί αυτή η μέθοδο. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτή την μέθοδο και να μην αφήσουμε τα πάντα στην Ολομέλη, διότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ξέρουμε ότι φεύγει από τον έλεγχο όχι μόνο των κοινοπτικών ομάδων, αλλά και των ίδιων των συμφερόντων τη Επιτροπή Αλία. ω εκ τούτου θεωρώ θα πρέπει να καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια, να χρησιμοποιήσουμε την ε, διαδικασία που προβλέπεται και αν μείνουν κάποια θέματα σε κρεμότητα για την Ολομέλεια, μπορούμε να τα συζητήσουμε και να δούμε τι τροπολογίε ε, από αυτέ που δεν έγιναν δεκτές μπορούμε να καταθέσουμε στην Ολομέλεια. Εγώ συμφωνώ να ε, ακολουθήσουμε την διαδικασία αυτή του άρθρου 50 και ελπίζουμε τα πράγματα να μπορέσουν να βελτιωθούν στο μέλλον. Κυρία Πατράου. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι ότι μπερδεύτηκαν κάπως οι συνάδελφοι γιατί έχουν λίγο χρόνο για τις τροπολογίες μέχρι αύριο το μεσημέρι όμως δεν μπορώ παρά να πιστήσω την προσοχή σας ε, για το ότι αυτή η ενισχυμένη συνεργασία ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ήταν δύσκολο να επιτευχθεί και ανοίγει ένα προηγούμενο σημαντικό για το μέλλον, όπως υπόθηκε. Για άλλες ε, περιπτώσεις ε, σκεφτόμαστε να διεκδικήσουμε και πάλι αυτό το καθεστώς της Ενδεδεμένης Επιτροπής και αν εμείς τώρα ζημιώσουμε αυτό που έχουμε πετύχει, δηλαδή μην προχωρώνται με τι τροπολογίε ή προτείνοντα οποιαδήποτε τροπολογία που δεν θα γίνει αποδεκτή γιατί θα είναι εκπρόθεσμη, τότε τελικά θα παραποδίσουμε μια σημαντική διαδικασία. Εγώ αναγνωρίζω ότι είναι λίγος ο χρόνος, όμως εδώ διακυβεύονται πολλά. Πέραν αυτού, ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να μιλάμε Έχω αρχίσει εγώ να συνομιλώ με την Επιτροπή Μεταφορών. Μία πτυχή που πάντοτε τεθώ πρώτη είναι ότι είναι και το κοινό μας ε, έργο ε, θα δημιουργούσε χρονικά προβλήματα. Αυτό μου έλεγαν από την πρώτη στιγμή, ότι θα καθυστερούσαν οι εργασίες. Εγώ δεν ε, ήθελα να τους δώσω ε, λόγο να δικαιωθούν ήθελα να σεβαστώ τις προθεσμίες και δεν ήθελα σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσω κανένα εμπόδιο κανένα πρόβλημα που θα μπορούσε να το επικληθούν εναντίον μας στο μέλλον. Να το επικαλεστούν εναντίον μας στο μέλλον όταν θα, όταν θα ξαναζητούσαμε την ενισχυμένη συνεργασία. Ξέρω ότι σας ζητώ να κάνετε μία θυσία, αλλά θα σας ε, καλούσα να κάνετε κάθε δυνατή προσπαθία να καταθέσετε στις τροπολογίες αύριο το μεσημέρι και να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν ε, πιο ρευστή αυτή τη διαδικασία γιατί δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ένα προηγούμενο για, τα, για τις μελλοντικέ εκθέσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πατράου. Μόνο ένα συνάδελφο προτείνει να ακολουθήσουμε την ε, διαφορετική διαδικασία. Η πλειοψηφία είναι υπέρ τη ε, διαδικασίας ε, που σας παρουσίασα. Έτσι διατηρώ την πρόταση που διατύπωσα. Να πω στον κύριο Αρσένη ότι αυτά τα συζήτησαν οι πολιτικές ομάδες. Εάν εσείς δεν έχετε προφόρηση, λυπάμαι, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό το έχουν αποφασίσει οι πολιτικέ ομάδε. Τώρα δεν ξέρω αν ε, υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην ενημέρωση βουλευτών από πλευράς πολιτικών ομάδων. Δεν ευθύνομαι. Νομίζω πως ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της μεσίας διατάξεως ε, και περνάμε στο επόμενο που είναι το πρωτόκολλο Συμφωνίας Ελευτικής Σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον και των ομόσπονδων πολιτιών της Μικρονησίας. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου. Una señalé, alors si se señalé. Bueno, a ver, eh, este acuerdo de. Αυτή η αλληλευτική συμφωνία στην προηγούμενη συνεδρίαση σας ε, ενημέρωσα ήδη και μια που όλα αυτά φαίνονται στην ε, έκθεση που έχω συντάξει έχει διανεμηθεί, δεν έχει διανεμηθεί η έκθεσή μου. Ναι. Έχετε γραπτός λοιπόν όλα όσα είχα πει την προηγούμενη φορά. Δεν θα χρειαστεί λοιπόν να στα επαναλάβω συνοψίζοντας να πω ότι πρόκειται για μια ανανέωση ενός πρωτοκόλου που ήδη ισχύει. το πρωτόκολλο για τους λόγους που σας εξήγησα την προηγούμενη φορά που είναι ίσονο σημασίας. Για λόγους ίσονο σημασίας δεν μπορέσε να δεν μπορούσε να προχωρήσει χρηματική αντιπαροχή για ένα παράδοξο ζήτημα ότι δεν είχε λογαριασμού σε ευρώ ή μικρονησία και έτσι δεν μπορούσαν να καταβληθούν τα ποσά και ω εκ τούτου κατεβλήθη το πρώτο κομμάτι τη χρηματική περιπτωροχής και οι πλειοκτήτες ε, κατέθεσαν τη δική τους ε, συνεισφορά δεν μπορέσαν λοιπόν να καταβληθούν τα ποσά και έτσι δεν εξετελέστη η προηγούμενη συμφωνία. Κατατέθη η πρώτη δόση και από τους ε, πλειοκτήτες ε, η ανανέωση λοιπόν ε, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε στο παρελθόν του Βουλγού Πετρόκολλο και αυτό το οποίο κατέστη σαφές αυτή τη φορά είναι ότι η χρηματική αντιπαροχή που κατέθεσε η Κομισιόν θα αφαιρεθεί από τις καταβολές των επόμενων χρόνων, άρα δεν θα πρόσουμε δύο φορές το ποσό. Το ίδιο συμβεί και με τις άδειες ε, για τις οποίες ήδη έχουν πληρώσει οι πλειοκτήτες, ε, οι ε, Έχουμε και κάποιες άλλες συμφωνίες ό,τι φορά το Μπάτι και την ίσους του Σολομόντα. Η Κομισιόν λοιπόν αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι ε, ότι επειδή υπάρχουν μια σειρά από συμφωνίες γνωρίζετε ότι εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ λίγα αλληλευτικά σκάφη αν δεν κάνω λάθος ε, τέσσερα γρηγρή και επτά παραγαδιάρικα η παρουσία μας λοιπόν όπως καταλαβαίνετε είναι ελάχιστη στην περιοχή και μετά από τα όσα σας ε, είπα, σχετικά με τα όσα συνέβησαν στον οργανισμό ε, αλληλείας του Δυτικού Κεντρικού Ειρηνικού, η παρουσία αυτή την περιοχή, όχι μόνο των αλληλευτικών σκαφών, αλλά και τη παρουσίας μας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και των συμφωνιών γενικότερα, αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας ωφελήσει είναι ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια για μεγαλύτερη ε, αηφορία των πόρων. Είναι η πλουσιότερη σε αλληλευτική περιοχή της ε, Φιλίου αυτή, ε, μία από τις πλουσιότερες και η κατάσταση των πόρων εξακολουθεί να είναι γενικά καλά καλή, αλλά υπάρχει το πρόβλημα της ε, παράνομης και λαθρέας και άναρχης αλίας και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τις χώρες αυτές, να εφαρμόσουν μια πολιτική διατήρηση των πόρων. Το πρόβλημα είναι ότι προτιμούν να έρχονται σε συμφωνία με την Κίνα παρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. και με λίγα λόγια οι μόσπονε πολίτε Μακρονησίου δεν ε, επιθυμούσαν να συνάψουν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με την Κίνα διότι η Κίνα έχει κάποιους ε, κανόνες ε, διατήρησης των πόρων που δεν είναι τόσο αυστηρές θα έλεγα όσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο χαλαρές αυτές οι ρυθμίσεις ως εκ τούτου λοιπόν θεωρώ πως ε, για αυτούς τους λόγους που προανέφερα, πρέπει να υπάρξει όλο και πιο μια μεγαλύτερη εγκατάσταση αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια παρουσία της Ευρωπαϊκής στην περιοχή ώστε να μην ε, διολυστήσει η κατάσταση. Νομίζω πως ε, αυτή είναι μια συμφωνία ίσονος σημασίας και τα ποσά δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε τέτοιου είδου συμφωνίε και τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν ε, έχουν επιληθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον μου το διαβεβαίωσε. Προτού να δώσω το λόγο στον κύριο Λαβάνια και κύριο Αρσέν, να κάνω μια ερώτηση προ την Επιτροπή που είχε μείνει αναπάτη την περασμένη φορά. Η Κομισιόν μου εξήγησε πως στα ε, τέλη Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο των ε, πολιτείων της Μικρονησίας ε, θα προκειμένου να εγκρίνει αυτήν την ε, συμφωνία και θα ήθελα να μάθω εάν δόθηκε το καλός έχει από το Κοινοβούλιο των Πολιτείων της Μικρονησίας. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Καντέκ και μετά ο συνάδελφος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η υπογραφή το 2006 και η εξέταση από τότε μέχρι σήμερα μας έδειξε ότι τίποτα δεν έχει τηρηθεί. Κανένα από τους τέσσερις γρήγοροι που ζήτησαν άδεια δεν την έλαβαν, δεν υπήρξαν ε, ε, παρόλο που υπευλήθη το ποσό, το χρηματικό, απολύτως καμία ποσότητα αλληλμάτων. Θέλουμε λοιπόν εδώ αυτό να λυθεί με σαφήνεια. Όσον αφορά την αλληλεία PLA, θα πρέπει να πούμε ότι βεβαίως πρέπει να παραμείνουμε στην περιοχή, να ενισχύσουμε την παρουσία μας, την παρουσία της ε, κοινότητας και παρόλο που οι ποσότητες που ελεύονται είναι σωστές, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε να γνωρίσουμε αυτόν τον τομέα της αλληλείας ε, πλά. Πρέπει βεβαίως να τηρηθούν ε, οι ποσότητες, αλλά είναι απαραίτητο να συμμετέχουν εδώ και άλλες χώρες. Ήμασταν παρόντες σε μια συνάντηση και το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης μας έδειξε ότι τα πράγματα είναι λίγο παράξενα εκεί πέρα. Βεβαίω θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να τηρηθεί αυτό το πρωτόκολλο και να υπάρχει παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις μικτές επιτροπές. Ευχαριστώ. Κυρία Λουή. Ευχαριστώ πολύ. Ως εισηγήτρια μας παρουσιάσατε εδώ κάποιες σαφείς δηλώσεις, τσεκτιμπό. εκτιμώ σε ό,τι αφορά την παρουσία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, στη σχετική περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης αλίας και καθώς αποτελεί και το παράδειγμα, δεν είναι το παράδειγμα σε αυτή την περιοχή, επί της αρχής συμφωνώ όμως, είπατε, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά το πώς έχει εφαρμοστεί η συμφωνία μέχρι σήμερα. Καταρχήν, για το καθεστώς των ενδιαφερομένων αποθεμάτων. Είναι αλήθεια ότι εξακολουθούμε ε, ε, να αλλιεύουμε εκεί το τόνο. Ε, βέβαια η παλαμίδα δεν υπεραλλιεύεται, αλλά αν διαβάσουμε τα στοιχεία από την έκθεση βλέπουμε ότι ο κυτρινόπτερος τόνος έχει φτάσει μόνο το 30% της αναπαραγωγικής βιομάζας και των μη αλλιευμένων επιπέδων που είναι πολύ χαμηλό μεγαλόφθελμος τόνος υπεραλλιεύεται Βέβαια και θα πρέπει να μειωθεί η θνησιμότητα μεταξύ του 34% και του 50% ο ψηφία πιθανότητα δεν υπεραλλιεύεται, αλλά τα στοιχεία δεν είναι πολύ αξιόπιστα. Έχουμε λοιπόν έλλειψη δεδομένων ε, σε ό,τι αφορά τα παραλλιεύματα. Ε, υπάρχουν ε, πολλές ανησυχίες ότι πολλά θηλαστικά όπως φάλαινες, δελφίνια αλλιεύονται ως παραλλιεύματα. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν αν η Μικρονησία ε, συνεργάζεται με τα γειτονικά κράτη όπως ε, η Γουινέα, η Γουάμ και άλλα κράτη για να συντονίσει την ε, αλίευση αυτών των ειδών τα οποία είναι μεταναστευτικά και μετακινούνται σε αυτά τα είδατα. Η Μικρονησία θα έπρεπε να έχει προβεί σε ένα συντονισμό με τα κράτη αυτά αν μπορούμε εμείς ε, εδώ να θεωρήσουμε ότι είναι βιώσιμο το απόθεμα των ειδών αυτών σε αυτή την περιοχή. Επίσης ξέρουμε τι αλλιεύουν η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Κορέα σε αυτή την περιοχή. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε και αυτό ε, για να δούμε αν συνεισφέρουμε στην υπεραλίευση ή όχι. Και κάτι ακόμη. Ξέρω ότι ποτέ δεν εκδόθηκαν οι άδειε. Ε, Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα πρωτόκολλο μεταξύ Μικρονησίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σύμφωνα με την αξιολόγηση και συστήνω σε όλους να το διαβάσει, αυτό γιατί όταν ε, μιλάμε για την προσέγγιση εταιρικής σχέσης μεταξύ Μικρονησίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως πάντοτε συμβαίνει με τέτοιε συμφωνίες, ένα τμήμα των χρημάτων θα έπρεπε να έχουν ε, χρησιμοποιηθεί για την προώθηση υπεύθυνων ελευθερικών πρακτικών στη Μικρονησία και οι αξιολογήσεις δηλώνουν με σαφήνεια ότι κατά τη διάρκεια των ε, τριών πρώτων ετών καμία από αυτή τις ρήτρες δεν έγινε σεβαστή. Η κοινή δέσμευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Μικρονησίας ε, ποτέ δεν τέθηκε σε εφαρμογή και δεν υπήρξε ποτέ και αμοιβαία συμφωνημένο πολιετές πρόγραμμα ούτε διάλογος για την ελευτική πολιτική μεταξύ των δύο μέρων. Έτσι λοιπόν δεν ε, μπήκε σε διάλογο καθόλου η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Μικρονησία σε ό,τι αφορά την ελευτική πολιτική. Αυτό εξηγήθηκε εκ νέου και το αναγνωρίζω αυτό και από άλλες αξιολογήσεις. Ε, δηλαδή, γιατί αποδόθηκε ήταν ότι είναι πάρα πολύ μακριά αυτή η χώρα από την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, πολύ εύκολα στέλνουμε ελευτικά σκάφη στη Μικρονησία, αλλά δεν μπορούμε να στείλουμε κάποιον από τις Βρυξέλλες για να συνομιλήσει ε, με ε, του ηθήνοντες εκεί στη χώρα και αυτό είναι απαράδεκτο. Βρίσκουμε την ίδια εξήγηση και σε άλλες αξιολογήσεις ε, αυτών των συμφωνιών στον ειρηνικό και η σύστασή μας είναι ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται κάποιοι στην περιοχή αν θέλουμε να συνάπτουμε αλληλευτικές συμφωνίες με τόσο απομακρυσμένες χώρες θα πρέπει να έχουμε και το προσωπικό επιτόπου που θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτές τις ε, κοινέ συναντήσεις ε, και να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με σοβαρότητα προωθεί την υπεύθυνη αλληλεία και δεν ε, είναι μόνο όλα αυτά λόγια στο χαρτί. Συνοπτικά λέει η αξιολόγηση ότι μπορεί να συναχθεί ότι οι συνιστό εταιρική σχέση της συμφωνίας ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη. Επίσης προκύπτει ότι η εταιρική σχέση με τις άλλες νήσους, το Κυριμπάτι και τις νήσους Σολομόντα έχουν το ίδιο χαμηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά την επίδεξη των στόχων. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία για την ενίσχυση της ελευτικής υπεύθυνης αλευτικής πολιτικής των χωρών αυτών. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει εδώ να δείξουμε σοβαρότητα και επίσης αξιολόγηση ε, αναφέρεται και έχει να κάνει και με την αξιοπιστία μας έναντι ε, ε, άλλων εταίρων της Δυτικής Αφρικής γιατί το χάρη δεν δίνουμε χρήματα στη Μαυριτανία γιατί δεν έχει υλοποιήσει όσο υποσχέθηκε στην Λευτική Συμφωνία Σύμπριξης και δεν το πράττουμε στον Ειρηνικό. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί από αυτού και πρέπει να ζητήσω από την Κομισιό να μας εξηγήσει και πάλι πώς ε, δείξατε μια τέτοια στάση αμέλειας ε, σε ό,τι αφορά τον ελληνικό ωκεανό. Και κάτι ακόμη να προσθέσω. Σε ό,τι αφορά την ε, ταξινόμηση αυτών των αξιολογήσεων να προσθέσω Νομίζω ότι είναι σκανδαλώδες που εμείς τα μέλη αυτή της Επιτροπής ε, πρέπει να πάμε και να καθόμαστε σε μια αίθουσα στη γραμματεία για να το διαβάσουμε αυτό θα πρέπει να είναι διαβαθμισμένο το έγγραφο. Δηλαδή, αν δεν έχουμε εμεί πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας ε, ως ε, κλαγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Οι πολίτες μας ψήφισαν εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας και παρεμποδιζόμαστε γιατί δεν έχουμε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες και μάλιστα οι φορολογούμενοι έχουν πληρώσει για αυτέ τι αξιολογήσει και πληρώνουν οι φορολογούμενοι και για τι ελευθερικέ συμφωνίε. Είναι σκανδαλώδε λοιπόν που είναι διαβαθμισμένα τα έγγραφα αυτά. Eh, Ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο. Ευχαριστώ η έλλειψη του τόνου στον ειρηνικό είναι 2.500 ε, τόνου και θα έχουμε 8.000 τόνους. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν υπάρχει διαφοροποίηση όμως το 70% αυτές τις αλλιεύσεις του τόνου γίνεται σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και αν ε, θέλουμε να εστιάσουμε ε, στο να έχουμε μια υπεύθυνη πολιτική αλίας πρέπει να είμαστε παρόντες στην περιοχή γενικά. Η κατάσταση του παθέματος ε, του τόνου είναι καλή, είναι μεταναστευτικό είδο. Ε, έτσι λοιπόν ένα σύνολο συμφωνιών είναι σημαντικό. Αυτή είναι η τρίτη συμφωνία. Εμεί συμφωνούμε να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και για να προωθήσει την αηφόρο αλλά και για οικονομικού λόγου και πρέπει να αυξήσουμε την παρουσία μα εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό συμφωνούμε με το προσανατολισμό της εισηγήτριας, δηλαδή να εμπλέκεται περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία και συμφωνούμε με τις προτάσεις. Θεωρούμε ότι οι στόχοι της ε, συμφωνίας ε, του 2006 σε σχέση με το πρωτόκολλο που δεν χρησιμοποιήθηκε συνεχίζουν να ισχύουν δηλαδή να ε, αναπτύξουμε τον έλεγχο, να έχουμε προμήθεια της ε, κοινοτικής αγοράς, να έχουμε φοροελίες. Φυσικά εμείς λαμβάνουμε αυτά τα προϊόντα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εισαχθεί σε αυτήν την αγορά και αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ θετική για να το πράξουμε. Με πάσα επιφύλαξη βέβαια ε, που υπάρχει στην πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστώ κύριος ε, Στίβενσον. Πολύ σύντομα ένα σχόλιο. Συμφωνώ με την τελευταία παρατήρηση. Όμως, όπως είπε στα εισαγωγικά της σχόλια η πρόεδρος, συναντηθήκαμε την προηγούμενο καλοκαίρι με μια αντιπροσωπεία από την Μικρονησία και αυτά τα οποία αναφέρατε, έλλειψη επικοινωνίας, και οι πληροφορίες που δεν φτάνουν ως εκεί, η αντιπροσωπεία αυτή ήρθαν και μας ε, παραπονέθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν όσον αφορά τα πολύ χαμηλά ποσά αποζημιώσαν αντιπαροχή που τους πληρώνουμε. Ενώ τα ποσά που πληρώνονται για τις άδειες είναι τελείως διαφορετικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο, διότι φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη, αν θέλετε, σοβαρότητας ή, εν πάση περιπτώσει, αντιμετώπιση σοβαρής από μέρους της δικής τους κυβέρνησης. Και βλέπουμε τι γίνεται και στις σχέσεις με την Κίνα. Ενώ, λοιπόν, είναι καλό το ότι εμείς έχουμε κατά κάποιο τρόπο βάλει ένα πόδι σε αυτήν την περιοχή ο ρόλος της ασφάλειας, της βιωσιμότητας των αλληλευμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως εξάλλου και σε όλες τις περιοχές που είμαστε δραστηριοποιημένοι. Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Νομίζω ότι η Λομαντρίλη κάλυψε τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω. Γενικές αρχές όμως είναι αυτές που με απασχολούν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε κι εμείς να εξάγουμε τις αρχές μας, τις αξίες μας. Και αυτές οι αληθικές συμφωνίες μπορεί να είναι ένα μέσο για να κάνουμε ακριβώς αυτό, δηλαδή να εξάγουμε την εμπειρία μας για μια βιώσιμη αλληλεία. Και μέχρι τώρα το έχουμε αποτύχει αυτό, δεν το καταφέραμε. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν στηρίζουμε την αλληλευτική μας πολιτική στα πλεονάσματα αλληλευμάτων. Και βεβαίως έχουμε συμφωνίες με πολλές άλλες γειτονικέ περιοχές. Μιλάμε βεβαίως για άλλα είδη μεταναστευτικά είδη. Θα πρέπει όμως να έχουμε κοινέ συμφωνίες για αυτά τα είδη, έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα αυτή να διασφαλίσει την βιωσιμότητα αυτών των πόρων. Την ίδια ώρα, με διάφορες διασυνοριακές συμφωνίες, την ίδια ώρα θα πρέπει να είναι σαφής οι επιπτώσεις επί της ανάπτυξης. Δηλαδή, στέλνουμε κάποια ποσά τα οποία θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να απορροφηθούν. Θα ήθελα να θίξω και δύο σημεία. Το ένα το ανέφερε η Ιζαμπέλα. Είναι απαράδεκτο το θέμα της διαβάθμισης των εγγράφων. Εδώ πραγματικά δημιουργούνται δυσκολίες και εμπόδια στην επικοινωνία, στην πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα και πώς είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να φτάσει σε αυτή τη συμφωνία η οποία είναι προσωρινή και η οποία ουσιαστικά από το Φεβρουάριο του 2010 εδώ και ένα χρόνο εφαρμόζεται. Αυτό είναι απαράδεκτο να μην έχουμε ε, πρόσβαση, δεν είμαστε ε, μαριονέτες και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο βάσει της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Ο κύριος Μπέρκ από την Κομισιόν έχει λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ ε, την έκθεσή σας ε, που θεωρώ πως είναι πληρέστατη και ιδιαίτερα ενημερωτική για αυτή τη συμφωνία με την Μικρονησία και που λαμβάνει υπόψη της, τη σημασία της παρουσίας ε, του Ευρωπαϊκού Αλευτικού Στόλου στην περιοχή. Κάνετε μια πολύ σωστή περιγραφή, αντιμετωπίσαμε όρους σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή του προηγούμενου πρωτοκόλλου, αλλά εδώ και λίγο χρόνο λάβαμε κάποιες εγγυήσεις, εγγυήσεις ε, σχετικά με τις ε, τραπεζικές πληρωμές, ε, εγγυήσεις ώστε τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν και που δεν χρησιμοποιήθηκαν και άρα δεν χορηγήθηκαν άδειε θα μπορέσουν να αφαιρεθούν από το μελλοντικό πρωτόκολλο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο ιδιαίτερα σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία κύρωσης ε, από πλευράς ε, Μικρονησίας, υπήρξε ένα σχέδιο ψηφίσματος ε, που υπολήθηκε στο, στο Συμβούλιο της Πολυνησίας πέρυσι τον Ιούνιο. Αυτό δεν εγκρίθηκε, αλλά πρόκειται να εγκριθεί τις προσεχείς εβδομάδες μετά από την τελευταία συνεδρίαση εδώ στην Ευρωπαϊκή Αλβίας υπήρξε μια αλλαγή στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Αλία ε, τη Μικρονησία και ένα νέο Γενικό Διευθυντή υπεύθυνο για θέματα Αλία ε, ε, διορίστηκε στα μέσα Φεβρουαρίου. Ήρθαμε σε επαφή λοιπόν με τι αρχέ τη Μικρονησία και ελπίζουμε ότι τις προσεχείς μέρες ή εβδομάδες το Συμβούλιο της τη Μικρονησία θα κυρώσει τη συμφωνία τώρα. Πολλοί αναφερθήκαν ε, στην ε, παράνομη και λαθρέα ε, και αναρχιαλία. Είναι όντως ένα γεγονός το οποίο γνωρίζουμε το ε, μόνο μέσω μιας περιφερειακής προσέγγισης θα μπορέσει να επιλυθεί το θέμα. Ε, αυτό απαιτεί μια παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή που συχνά με δυσκολία ε, μπορεί να ε, ακουστεί η φωνή της. Τώρα επανέρχομαι στα αποθέματα που έθεσαν ε, διάφοροι ευρωβουλευτέ. Δύσκολα μπορούμε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα στη συμφωνία με την Μικρονησία, διότι δεν υιοθετήθηκε στην προηγούμενη περίοδο. Αλλά αν παρατηρήσουμε το τι συμβαίνει στι ε, νήσου του Σολομόντα, παρατηρούμε ότι περισσότερα αλλιεύματα τη περιοχή αφορούν το είδος ε, τόνου skipjack. Ε, θεωρούμε όμως ότι αυτό ε, ο αλευτικός σπόρος δεν τη χάνει Ε, υπάρχουν κάποιες μεγαλύτερες ανησυχίες αναφορικά με άλλα είδη τόνου όπως τον μεγαλό θαλμοτόνο ε, θα λαμβάνουμε σε αποφάσεις που είχαν ευθεί από την ε, Επιτροπή ε, διαχείριση των στην που προβλέπει την μείωση κατά 30% των ε, αλλιευμάτων των μεγαλόφθαλμου. Θα προσεχείρεται εφαρμόζονται. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτήν την ε, περίοδο. Παρατηρούμε λοιπόν την κατάσταση των αποθεμάτων. Η αληθή προσπάθεια έχει περιοριστεί την περίοδο αυτή και θεωρώ ότι όλα αυτά βρίσκονται σε ευθεία γραμμή με τις ανησυχίες μας σχετικά με την διατήρηση των πόρων. Επανέρχομαι τώρα στο ζήτημα της στήριξης ε, του κλάδου. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι δεν υπήρξε μεικτή επιτροπή κατά τη διάρκεια προηγούμενη συνάντηση. Οργανώθηκε μια τέτοια συνάντηση το Μάιο του 2010. Όντω η προηγούμενη συμφωνία δεν εφαρμόστηκε όσο έπρεπε και λυπούμεθα γι' αυτό. Αλλά τώρα Ας ανατενίσουμε το μέλλον. Έχουμε λάβει κάποιες ε, ε, ρυθμίσει ε, για την σωστή εφαρμογή. Υπάρχει μια ρήτρα που μας επιτρέπει την διακοπή της εφαρμογής εάν δεν γίνεται με τρόπο σωστό. Μικτή Επιτροπή θα συνέλθει τους προσεχείς μήνες, προ... πιθανότατα τον Απρίλιο, το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί και αυτή η μεικτή επιτροπή που θα είναι η πρώτη που θα συνεδριάσει υπό το νέο πρωτόκολλο θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της κλαδικής στήριξης και θα πρέπει να οδηγήσει στη συμφωνία ειδικά με μια μήτρα θα λέγαμε ε, παρακολούθησης ε, τη καταστάσεω στην Μικρονησία. Τώρα ε, το θέμα τη παρουσίας μας στον Ειρηνικό είναι κάτι που τονίστηκε. απόσπαση ενό εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενό διαπιστευμένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε, μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στα σκαριά, αλλά η δημιουργία μιας τέτοιας θέσης διαπιστευμένου αιματαλίας είναι γεγονός πλέον. Τώρα το ζήτημα της αξιολόγησης και το χαρακτήρα ο διαβαθμισμένος αυτής της έκθεσης το σημειώνω αυτές τις παρατηρήσεις ε, που ακούστηκαν. Θεωρώ ότι το ζήτημα ξεπερνάει το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και χρειάζεται να αναφερθεί στους ανωτέρους μας ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, κάποια θέματα διαδικασίας. Τώρα, η τελευταία αξιολόγηση post ε, που λάβαμε και δεν είναι διαβαθμισμένη είναι ακριβώ για τη Μικρονησία. Τώρα από εκεί και πέρα άλλαξαν τα πράγματα, πράγμα το οποίο το τόνισα εγώ και μου φαίνεται παράλογο. Όμω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανεί δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει γιατί ακριβώς ε, εγώ πιθύνθηκα στον κύριο Σέρσκοβιτς και δεν κατάλαβα τι του έλεγα, αλλά από τον Ιούνιο εκθέσεις που έφταναν ε, αρχικά στο Κοινοβούλιο ελεύθερα, ξαφνικά έγιναν εμπιστευτικά έγγραφα. Έτσι λοιπόν εγώ θα προτείνω στους συντονιστές από εδώ και πέρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που προβλέπετε στην Διοργανική Συμφωνία Πλαίσιο να αμφισβητήσουμε αυτές οι εκθέσεις εξ προσταξιολόγησης να είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, να είναι διαβασμένες γιατί δεν σέβονται τα κριτήρια της Διοργανικής Συμφωνίας Πλαισίου και επίσης ε, έχουμε και ένα προηγούμενο και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα Απλώς ε, ξαφνικά άρχισαν τα έγγραφα να μετατρέπονται σε διαβαθμισμένα έγγραφα. Ξέρετε, αυτές οι εκθέσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ε, για τη δουλειά μας, είναι τεχνικού χαρακτήρα, επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι διαβαθμισμένα. Και προτάθηκε εδώ από τη συνάδελφο ο κανόνα να είναι να μην είναι εμπιστευτικά τα γραφεία αυτά, εκτό από ορισμένε περιπτώσει, γιατί μπορεί, παραδείγματο χάρη, να είναι πιο ευαίσθητα έγγραφα αυτά από πολιτική σκοπιά σε ορισμένε περιπτώσει. Μέχρι τώρα, βέβαια, δεν έχω λάβει απάντηση. Λοιπόν, πάντως ε, μην ανησυχείτε, έχουμε και το άρθρο 50 και νομίζω ότι είναι λογική η θέση μας ε, και νομίζω ότι δεν ε, είναι σωστή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, για το δεύτερο θέμα διαδικασία, το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Σερσένη, ήδη έχουμε καταρτήσει μια διαδικασία Υπάρχει μια συμφωνία με τη Μαυριτανία για το μέλλον και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε σε τριμηνέα βάση να μας στέλνουν λεπτομερή στοιχεία για το ε, ποιες πιθανές οδηγίες μπορεί να είναι υποδεπραγμάτευση έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένο το Κοινοβούλιο από την αρχή των διαπραγματεύσεων στα θέματα που θεωρούμε εμείς σημαντικά γιατί ξέρετε ότι δεν είναι και εύκολο να κάνουμε μια εξαιρετική διαδικασία, πρέπει να επιλέξουμε. Όμως ε, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με τη Μαυριτανία, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και θα δούμε και πώς θα το αξιολογήσουν και οι βουλευτές. Γιατί κατόπιν πρέπει να θέτουμε σε εφαρμογή όλα συζητάμε και να παρευρισκόμαστε στις μικτές επιτροπές και τα λοιπά. Ξέρετε, είναι πολλή δουλειά. Τώρα, πέραν αυτών, να αναφερθώ στη συμφωνία με τη Μικρονησία να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπόρεσε να γίνει καμία αξιολόγηση της τομέκης στήριξη, ε, γιατί δεν τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία. Δηλαδή πληρώθηκε η συμφωνία αυτή αλλά δεν υπήρξε εκτέλεση ή εφαρμογή αυτής. Όμως εγώ αυτό που θέλω να ξεκαθαριστεί εδώ γιατί μου φαίνεται ότι είναι πιο ξεκάθαρη ιδέα είναι το εξής οι Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας, όπως ε, και πολλά άλλα κράτη του δικοκεντρικού Ειρηνικού, συμμετέχουν σε μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης αλίας, η οποία λειτουργεί αρκετά άσχημα ήδη. Και Μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή έχει διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά μειοψηφικό με άλλες χώρες. Ε, είμαστε πάντοτε σε μειοψηφική θέση σε σχέση με άλλες νησιωτικές χώρες ε, που έχουν ε, κάποιες θέσεις οι οποίες δεν είναι και ιδιαίτερα βιώσιμες ή εφόρες. Δηλαδή, αντιτάχθηκαν ε, καταρχήν στο ε, ε, υπάρχουν ε, τα μέτρα ε, του συστήματος για τα αλλιεύματα. Δεύτερον, στην Επιτροπή Αλλίας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού, όπως γνωρίζω, είναι η μόνη πόδα όπου εγώ είδα ότι πέρα από ε, τον καθορισμό της ε, ζώνης εφαρμογής ε, της σύμβασης υπάρχει τόσο μεγάλη εμπλοκή με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες δηλαδή ε, τα μέτρα που υιοθετούνται για τα μεταναστευτικά είδη κανονικά πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή. Όμως, από ερμηνεύεται η ίδια συμφωνία και τα μέτρα εφαρμόζονται μόνο στην ανοιχτή θάλασσα και όχι στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και με την ιδιαιτερότητα σε αυτή τη ζώνη του ειρηνικού το 90% σχεδόν είναι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Έτσι λοιπόν εγώ θέλω να τονίσω τη σημασία ε, να παρευρίσκεται εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να προσπαθήσει σε αυτές τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες να γίνεται σεβαστή η ευρωπαϊκή θέση έναντι των Κινέζων και των λοιπόν που βρίσκονται εκεί. Γιατί κανεί δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά είναι πολύ πιο βιώσιμε, όσοι και αν κάποιοι το αμφισβητούν. Ε, οι δικέ μα θέσει είναι καλύτερε από τη Κίνα ή των υπολείπων. Επίσης, ε, οι χώρες αυτές είναι ομαδοποιημένες ε, σε ε, διάφορα υποπεριφερειακά βήματα, σε διάφορα τέτοια φόρα. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να τονίσω εδώ πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μία φωνή που να υπερασπίζει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιστεύω ότι είναι σημαντικό στα θέματα αυτά να συμμετέχουμε, ακόμη και αν έχουμε 4-5 σκάφη. Βλέπετε ότι είναι ισχνή η παρουσία μας, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να μπορούμε να ελέγχουμε τη διαδικασία. Εδώ ίσως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ε, υποστήριξη στο να καλέσουμε ε, τους υπευθύνους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι επιτόπου εκεί για να ελέγχουν ε, την διαδικασία. Είναι σημαντικό κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια ζώνη του ειρηνικού που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά το Κυριμπάτι, παραδείγματο χάρη, αλλά από τι χώρε με, έχουμε, με την οποία έχουμε αλληλευτική συμφωνία, έχει τόσα πολλά νησιά το ίδιο το Κυριμπάτι που ε, μία φορά συνεδριάζει το κοινοβουλίο του. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν όλοι αυτοί από τόσα νησιά. Πάρα πολλοί ε, κόσμος δηλαδή, διασκορπισμένος. Υπάρχει δηλαδή γεωγραφική δυσκολία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι ε, πρέπει να λέμε και λέγεται στην έκθεση ότι πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Αν και βέβαια μπορώ να σας πω ότι έχει ασκηθεί πολύ μεγάλη κριτική στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με άλλες συμφωνίες, όμως εδώ ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί μπορώ να σας πω ότι είχαμε μειοψηφική θέση κυρίως όταν ε, αναφερόμαστε στο τι κάνουν οι υπόλοιποι σε σχέση με την ε, παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι ακόμη. Κυρία Μπιλμπάου. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη γιατί με κάλεσαν ακριβώς ε, τη στιγμή που συζητήθηκε η έκθεση αυτή. Εγώ θέλω να σα πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την έκθεσή σας. Είναι θέματα που έχουμε συζητήσει σε αυτή την Επιτροπή. Και ε, φυσικά είμαι υπέρ στο να προσυπογράφουμε όλες αυτές τις συμφωνίες και μπορώ να σας πω ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί να συνεισφέρει στο μέτρο του δυνατού στο να υπάρχει μια εφόρο αλία. Απλώ αυτό ήθελα να πω. Αυτή είναι η θέση τη ομάδα μου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας πω λοιπόν ότι 21 Μαρτίου είναι προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Από πού έρχεται αυτός ο θόρυβος. Δεν ξέρουμε από πού έρχεται ο θόρυβος αυτός. Λοιπόν, 29 Μαρτίου. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 12 Απριλίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή και θεωρητικά θα, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Μαΐου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το σημείο 7. Περάσουμε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξη, συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κρατός λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλληψη παράνομης λατρείας και άνορχης αλίας. Γνωρίζετε ήδη, σας το είπα και την περασμένη φορά, ότι εδώ απλώς ε, Μιλάμε για το εξιστιφάο το 2001 εκπονήθηκε ένα διεθνές σχέδιο δράσης ε, κατά της Ελίας Πλά, παράνομες ελευθερές και άναρχης Αλίας. Επίσης, ε, ο ΦΑΟ το 2005 έκρινε Ξέρετε ότι οι δύο κύριοι πυλώνε για την καταπολέμηση της ελία πλά είναι ακριβώς τα μέτρα του κράτους λιμένα και το σύστημα τεκμηρίωσης των ελευμάτων, ακριβώ αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Αυτοί οι δύο πυλώνες ε, είναι μάλλον ανήκουν στο σύστημα που ε, ενέκρινε φάω το 2005, ενέκρινε ορισμένα μέτρα κράτος λιμένα Ορίσαμε ένα ελάχιστο σύνολο μέτρων ε, που ήταν εθελοντικού χαρακτήρα και κατόπιν το 2007 η Επιτροπή Αλίας της ΦΑΟ εκπώνησε ένα δεσμευτικό εργαλείο που ολοκληρώθηκε το 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το επέγραψε φέτος το Νοέμβριο και τώρα αυτό που προτείνουμε είναι να συστήνουμε την έγκριση της συμφωνίας ε, σύμφωνα με το άρθρα 43 και 218 της συνθήκης. Λοιπόν, καλό είναι αυτό να το υπογράψουμε για να έχει τον ελάχιστο αριθμό υπογραφών. Δύο χώρες έχουν υπογράψει, νομίζω η Σιλάνκα και η Βερμανία μέχρι τώρα και χρειάζεται να συλλέξει ελάχιστο αριθμό χωρών για να τεθεί σε όμως, οποιαδήποτε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το υπογράψει, θα εγκριθεί. Αλλά θέλω να πω ότι τα περισσότερα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο του ΣΦΕΟΥ ήδη συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για την καταπολέμηση της Αλίας Πλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει στην ομοθεσία της τα μέτρα αυτά έτσι λοιπόν, ε, απλά πρέπει να εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα που θα είναι δεσμευτικό για όλους. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσες υπογραφές χρειάζονται, αλλά μόνο Σρι Λάγκα και Βερμανία έχουν υπογράψει μέχρι τώρα. Περί αυτού πρόκειται. Η συστασή μου λοιπόν είναι να πούμε ότι ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό για το θέμα αυτό. Όπως και να έχει η Επιτροπή ήδη το έχει συμπεριλάβει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την καταπολέμηση της ελίας πλά, όπως σας είπε ο κ. Στίβενσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τις συστάσεις που υποβάλλεται και όντως ε, η δικτή ομάδα ασχολήθηκε με το θέμα αυτής της παράνομης αλίας που πολλές φορές ήταν την εγκληματική δραστηριότητα. Πολλοί συμμετέχοντες είπαν ότι ναι, πολλές φορές είναι παράνομη, είναι μάλλον λαθρέα, αλλά δεν είναι πάντα παράνομη. Και όταν υπάρχουν κάποιες εγκληματικές συνέπειες, και αν λάβουμε υπόψη μας ε, τα δισεκατομμύρια στα οποία αφορά αυτά τα κλεμμένα αν θέλετε από θέματα, αλλιεύματα και θυμάμαι πολύ καλά τις προτάσεις της Επιτροπής που έλεγαν ότι είναι πολύ περήφανοι γιατί έχει υπογραφεί από ένα μεγάλο αριθμό χωρών το νέο, η νέα συμφωνία. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα στην πράξη. Αν μπορούσαμε ή τουλάχιστον να μπορούσαμε τουλάχιστον να τους κατονομάσουμε θα είχε γίνει μια συγκεκριμένη πρόοδος. Σήμερα τα αλλιευτικά σκάφη τα οποία επί χρόνια δρούν με αυτόν τον παράνομο λαθρέο τρόπο και αλλιεύουν, κατόπιν ε, μεταβιβάζουν σε ένα άλλο αλλιευτικό σκάφος ε, τα αλλιεύματα. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει εδώ μία εμπλοκή της παράνομης αλλά και της νόμιμης ε, αλλιευτικής δραστηριότητας. Και όλες, όλα αυτά φαίνονται στην έκθεση. Το ζητούμενο βεβαίω είναι τελικά τι ακριβώς ποσότητα αλλιεύτηκε. Και δεν μπορούμε να πούμε απλά και μόνο ότι πρόκειται για μια μεγάλη εγκληματική δραστηριότητα. Ε, δεν έχουμε κάνει απολύτως καμιά πρόοδο επί της ουσίας. Κοιτάξτε. Νομίζω πως ε, με τον κανονισμό πλά του 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όχι μόνο τη δυνατότητα, αλλά την υποχρέωση να απαγορεύσει τις εισαγωγές από χώρες που δεν εφαρμόζουν αυτούς τους βασικούς κανόνες. Τα μέτρα σε ό,τι αφορά το λιμένα κλπ. Υπάρχει νομική βάση και πολλές χώρες δεν το πράττουν. Αλλά χορηγούνται πιστοποιητικά στις χώρες αυτές προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντα τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, ποιος είναι η περιότητα του κυρίου Ντεγκούχ. Πάντως σύμφωνα με τον κανονισμό του 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απαγορεύσει τις εισαγωγές και αυτό το οποίο τις πονάει τις χώρες αυτές είναι οι εξαγωγές ακριβώς και η αδυναμία να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν ε, να... Όλες αυτές οι χώρες ε, του ειρηνικού όλοι είναι κατά του κάτι Documentation Scheme και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους έχει απειλήσει ότι θα τους αφαιρέσει τα πιστοποιητικά αυτά αλλά γιατί δεν το πράττει εντάξει ε, μπορεί να είναι αναπτυσσόμενες χώρες και δεν ξέρω εγώ τι, όλες αυτές οι ανοησίες. Υπάρχει ο κανονισμός, υπάρχει νομοθεσία και πρέπει να εφαρμοστεί και τους ασθένους. Ναι. ναι, φυσικά όπως είπατε. Θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτό την συμφωνία διότι είναι σημαντική για μας, αλλά είναι σημαντικό όλες οι χώρες ανά τον κόσμο να υιοθετήσουν αυτούς τους ε, κανόνες. Φυσικά ε, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε να υπογράψουν, αλλά θα πρέπει να λάβουν μέτρα που πηγαίνουν προς την αυτή κατεύθυνση. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, όπως είπατε, Πρόεδρε, αυτό ξεκίνησε από το ΦΑΟ του 2001, όταν ξεκίνησε να συζητάνε το ζήτημα της ΠΛΑ, άρχισαν να προετοιμάζουν τη συμφωνία και έχουμε τώρα την ε, δυνατότητα να συμφωνήσουμε. Γιατί επίση υπάρχει το θέμα ότι εδώ πρόκειται για τη μεγαλύτερη απειλή στην ε, βιώσιμη αλληλεία είπατε ότι το 20% των αλλιευμάτων που πολλούνται ανά τον κόσμο προέρχονται από αλλία πλά. Ένα δις ε, ευρώ είναι το κόστος αυτών των ε, ηχθείων που εισάγουμε. Γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα μέτρα του κράτους λιμένα, διότι είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί στις ανοιχτές θάλασσες η πλά, αλλά στα λιμάνια είναι πολύ πιο εύκολο να σκηθεί έλεγχος Τώρα να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία που προτείνει ο κανονισμός, το ζήτημα των ε, λιμένων, η χώρα κράτους, ε, μάλλον το κράτος λιμένα, το ρόλο των κρατών συγγνώμη, σημαία, του μηχανισμού διασφάλιση, του μηχανισμού ανταλλαγή προφοριών και όλα, αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ. Κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως είμαι υπέρ αυτής της πρότασης ε, συμφωνίας. Πρόκειται όμως απλώς για μια συμφωνία υπογεγραμμένη από πολύ λίγα κράτη. Είπαν και άλλοι συνάδελφοι εξάλλου ότι αυτή η παράνομη λαθρέα αναρχελία είναι παράνομη, είναι έγκλημα. Υπάρχουν μεγάλα κράτη τα οποία συμμετέχουν, όπως η Κίνα παραδείγματος χάρη, μην νομίζετε ότι έχω έμονη ιδέα με την Κίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι οι Κινέζοι ψαρεύουν παντού στον κόσμο και εμείς επιβάλλουμε στους δικούς μας αλείς και πλειοτήτες πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να επιβληθεί και να επεκταθεί αυτή η ρύθμιση. Ο ΠΟΕ, ο Πασκάλ Λαμή και άλλοι, αγνοούν πλήρω όλα αυτά και τους κανόνε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι ελεύθερε συναλλαγέ. Είμαστε φιλελεύθεροι, αλλά το να είναι κάποιο φιλελεύθερος σημαίνει ότι είναι υπέρ της ελευθερίας και όχι υπέρ της ζούγκλας. Αυτοί οι άνθρωποι μας εμποδίζουν να ρυθμίσουμε αυτήν την παράνομη αλία. Και ξέρετε πολύ καλά ε, από τη στιγμή που έχω υποβάλει την έκθεσή μου για τις αγωγές τι πιστεύω, ποιε είναι οι απόψει μου. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτήν την ε, παράνομη λαθρεαλία γιατί αυτό είναι που υπονομεύει όλο το σύστημά μας. Έχουμε επαγγελματίες αλείς, τους υποχρεώνουμε να τηρήσουν κανόνες για το περιβάλλον, υγειονομικούς κανόνες, κοινωνικούς. Όλοι αυτοί όμως δεν ε, σέβονται τίποτα ούτε τις ανθρώπινες ζωές και φυσικά ε, ούτε ε, τα αποθέματα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Ευχαριστώ κύριε Λόι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την εκθεσή σας. Φυσικά υποστηρίζουμε πλήρως ε, το να συμπεριληφθούν τα μέτρα κρατούς λιμένα στην κοινωτική νομοθεσία. Αργότερα θα αναφερθώ στο ΦΑΟ και στις σχετικές εμπειρίες μου. Όμως είναι κάπως απαθαρρυντικό να βλέπουμε το χαμηλό επίπεδο δέσμευσης ε, πολλών κρατών παγκοσμίω. Και όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, Πολύ λίγα έχουν υπογράψει μέχρι τώρα ε, τη συμφωνία για τα μέτρα κράτους λιμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε κάθε επίπεδο για να προσπαθήσει να πείσει και άλλα κράτη να προσυπογράψουν. Επίσης, ε, στο πλαίσιο και των αλευτικών ε, συμφωνιών, των συμφωνιών εταιρικής σχέσης είναι ένας από τους ε, πλέον αποτελεσματικούς τρόπους όπως το κόστος για να καταπολεμήσουμε την παράνομη ηλία παγκοσμίω. Ευχαριστώ και τον κύριο Στίβενσον που οργάνωσε το σεμινάριο για την ηλία πλά ως οργανωμένο έγκλημα. Είναι ένα θέμα που τέθηκε από την Ορβηγική κυβέρνηση καταρχήν αλλά το να ε, θεωρηθεί να κατηγοριοποιηθεί ως έγκλημα η άλλη απλά μας δίνει άλλα εργαλεία, άλλα μέσα για την καταπολέμηση αυτή τη αλία σε διεθνέ επίπεδο. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασία και με το ε, γραφείο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και του εγκλήματος ε, πέρα από το ΦΑΟ. Ε, Ένα εκπρόσωπο από το ΦΑΟ είπε ότι ο όρος crime, εγκλήμα ποτέ δεν ε, εμφανίζεται σε κανένα έγγραφο που να έχει να κάνει με την άλλη απλά. Έτσι λοιπόν θεωρείται περισσότερο διοικητικό αδίκημα παρά έγκλημα. Όμως Ξέρετε ότι έχουμε εδώ και φόρο διαφυγή με αυτές τις πρακτικές. Έχουμε ψευδείς δηλώσεις και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν εμπίπτει ε, σε μια σειρά ποινικών ε, νόμων. Δηλαδή θα ήταν ένας καλός τρόπος να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε έτσι σε αυτό το πλαίσιο την ε, παράνομη λαθρεία και αναρχιαλία και αυτό έχει συζητηθεί και από τις ΗΠΑ, την Ορβηγία και άλλες χώρες. Και νομίζω ότι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει συμφέρον να συμμετάσχει για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και με άλλα μέσα πέρα των μέσων που μας δίνει ο ΦΑΟ. Ο κύριος Σάντσες. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Απλώς ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ μας ακούστηκαν. Εγώ νομίζω ότι να έχουμε ένα διεθνέ πρότυπο για το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν είναι το ίδιο να υπερασπίζει κανεί μια θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να προσπαθεί να την επιβάλλει και στα υπόλοιπα κράτη. Ενώ αν έχουμε ένα διεθνέ πρότυπο, αποκτούμε μεγαλύτερη νομιμοποίηση και φυσικά μπορεί αυτό να ληφθεί υπόψη και στι συμφωνίε με τι τρίτε χώρε. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα μπορούσε να διευκολύνει πάρα πολύ την εργασία μα στον λόγο το με Ευχαριστούμε. Αγύρα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την εισηγητρία την εξαιρετική έκθεση που παρουσίασε για την ε, συμφωνία για τα κράτη λιμένα, όπως ε, σας είπα, εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεγράφει αυτή η συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο της κύρωσης, η Σρι Λάνκα και η Μιανμάρ, η έχουν υπογράψει. Χρειάζονται ακόμα 23 κυρώσεις για να τήθει σε ισχύ. Σε σχέση με όλη την πολιτική καταπολέμηση τη Ελία Πλάτ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία ένα θεμελιώδη πυλώνα ε, είναι ο κανονισμό Ελία Πλά που τέθηκε σε ισχύ 1η Ιανουαρίου του 2010, πρέπει να πούμε ότι η Κομισιόν ε, δεν έχει ε, καταβάλει την ε, ε, προσπάθεια, την τεράστια προσπάθεια για την εκπόνηση του κονισμού για να μην τον εφαρμόσει στη συνέχεια. Έκανε τεράστια προσπάθεια η Κομισιόν για να καταπολεμήσει ακριβώς αυτή την παράνομη αλία και εφαρμόζει αυτό το κανονισμό σε όλες τις πτυχές του, έτσι όπως προβλέπεται στο ίδιο το νομοθέτημα, με σταδιακό τρόπο και φυσικά θα εφαρμοστεί και θα υπάρξουν και κάποια εμπορικά μέτρα που εθετηθούν ακριβώς ε, για προϊόντα που εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από σκάφη με κοινωνικά, με, με ευρωπαϊκά με συμφέροντα που δεν φέρουν κοινοτική σημαία αλλά είναι κοινωνικών συμφερόντων. Ε, Τώρα, η συμφωνία αυτή θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να υποστηρίξουμε και να νομοποιήσουμε αυτές τις μονομερείς δράσεις που αναλαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του κανονισμού για την καταπολέμηση της ελίας πλά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε τη σημασία της κύρωσης αυτής της συμφωνίας που όπως σας είπα θα σημαίνει μια πολύ σοβαρή στήριξη για την νομιμοποίηση των δράσεων μας για την καταπολέμηση της ελίας πλά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και σας πρόεδρε αλλά και τους ε, υπόλοιπους ε, βουλευτές ε, για το έργο σας προκειμένου να καταλήξει σε καλό λιμένο αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να πω. Ο Φάου στις τελευταίες εκθέσεις και χαίρομαι που κυρία Ρωμέ ε, μας μίλησε περί αυτού και μπορεί να μας ε, αναφέρει και λεπτομέρειες ότι δεν ε, επιθυμούν να δεχθούν τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Ε, μιλάμε για ζώνες της Αμερικές που ονομάζονται αγγλιστή Creeping Jurisdiction και μια άλλη περιοχή είναι αυτή του Ειρηνικού. Υπάρχουν θέσει λοιπόν σαφείς που σχετίζονται με εθνικιστικές απόψεις και θέσεις. Πρόκειται λοιπόν για εθνικιστικές και υπερεθνικιστικές θέσεις που αφορούν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Το ζήτημα είναι κατά το μάλλον ή τον περίπλοκο Αυτά τα ζητήματα λοιπόν χρειάζεται να τα λάβει η Κομισιόν υπόψη της τα σοβαρά. Κάνουν κάποιες αξιολογήσεις ε, και όταν ε, θα έχουν τα αποτελέσματα πρέπει να μας ενημερώσουν και να ασκήσουμε πίεση στις χώρες αυτές. Ε, δεν αναφέρουμε τώρα στην και κλπ αλλά χρειάζεται κάποια στιγμή να μας πάρουν υπόψη τους οι χώρες αυτές. Τώρα για την κατάθεση τροπολογιών 21 Μαρτίου, το μεσημέρι προθεσμία 12 Απριλίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή και θα περάσουμε στην Ολομέλεια τον Μάιο. Περνάμε στο επόμενο σημείο της Διατάξεως που είναι το σημείο 10 είναι η συμφωνία με τις Σέιχελες. Ο κύριος Καντέκ είναι εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρουσίαση θα κάνω σύντομα όσον αφορά την ε, Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας των ΣΕΙΧΕΛΩΝ. Καλύπτουμε την ε, περίοδο από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του 2011 και πρέπει να ανανεώσουμε με κάποιες τροπολογίες, τροποποιήσεις που έχει διαπραγματευτεί η Επιτροπή αυτή τη συμφωνία. Βάσει της εντολής που έχει δοθεί από το Συμβούλιο, η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τις Σεϊχέλες για να ανανεώσει αυτήν την ε, συμφωνία. Ένα νέο πρωτόκολλο στις 3 ε, ε, Ιανουαρίου μονογράφηκε για τρία χρόνια. Πρόκειται για ένα αρχιπέλαγος με μια ζώνη οικονομικής ε, δραστηριότητας, μια παράκτη περιοχή που έχει πάνω από 1.350.000 χιλιόμετρα, μια πολύ σημαντική δηλαδή παράκτη περιοχή η Αλία δραστηριοποιεί 17% του πληθυσμού και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οικονομικό πόρο. 400 μονάδες αλληλευτικές, εκ των οποίων το 80% πρόκειται για παραγαδιάρικα επιφανείας. Όσον αφορά τώρα την αλία τόνου, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτών των αποθυμάτων, με 16,8 εκατομμύρια ευρώ για τα τρία έτη που καλύπτει το νέο πρωτόκολλο, 3,38 εκατομμύρια για 52.000 ε, τόνους ετησίως καθώς και το επιπλέον ποσό που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη της αλλιευτικής πολιτικής, της πολιτικής της Εχέλες, ένα ποσό των 2.220.000. Υπάρχει ένα σύνολο 60 σκαφών που αλλιεύουν κυρίως τρία είδη τόνου, 300.000 τόνοι το χρόνο. Το 2003 το, ε, η ποσότητα αυτή ξεπενούσε στους 4.000 τόνους. Βεβαίως σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια πειρατική δραστηριότητα που πλήττει τους ε, τοπικούς αλληλείς και έχει αυξηθεί και ο κίνδυνος της δραστηριότητας στην περιοχή αυτή. Όσον αφορά τα αλλιεύματα, 50% αφορούν την πρώτη ποιότητα τόνου, τόνος του Ινδικού ε, ωκεανού, με μια πλήρη εκμετάλλευση για τον τόνο τον κίτρινόπτερο Οι άλλες δύο κατηγορίες τόνου δεν εκμεταλλεύονται όσο θα μπορούσαν. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που δημιουργεί ανησυχίες με μια σημαντική μείωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τον γόνο του κοιτινόπτερου τόνου. Πρόκειται για μια ανεξέλεκτη δραστηριότητα από μέρους ε, ενός στόλου παράνομης λαθρέας άναρχης αλίας και για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την παράνομη αλία επιτρέπεται η δραστηριότητα μόνο σε σκάφη τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα σε δημόσια μητρώα ήδη από το 2003 έτσι ώστε να μην υπάρξει αυξανόμενη πίεση. Οι Σεχέλες έχουν επικυρώσει, έχουν υπογράψει τις περισσότερες διεθνείς συμφωνίες για το περιβάλλον και για την αλία και την διατήρηση των μέτρων ε, για την ανοιχτή θάλασσα. 30 θέσεις απασχόλησης, 760 στην Ευρώπη, για ε, δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα. Η αρχή για την αλληλεία των Σεϊχέλων είναι μία από τις πιο αρμόδιες, θα έλεγα, αρχές ε, στον τομέα της αλληλείας στον Ινδικό ωκεανό, που επιτρέπει να καταπολεμήσει την παράνομη και λαθρεαλία. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι τα αλληλευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και παρατηρητές ε, από την Ευρώπη αλλά και από την αρχή των Σεϊχελών. Χαιρετίζω σήμερα εδώ την παρουσία ενός εκπροσώπου της πρεσβείας των Σεϊχελών στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν λοιπόν κάθε φορά δύο άτομα από τις Σεϊχέλες ε, που βρίσκονται στον ε, κατάλογο που παρέχει ο πλειοκτήτης για τα άτομα που βρίσκονται επί των αλληλευτικών σκαφών. Δύο άτομα από τις αρχές αυτές των Σεχελών. Η Μικτή Επιτροπή δεσμεύεται σήμερα σε ένα πολιετές πρόγραμμα για την ε, βιώσιμη αλληλεία στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Δεύτερον, υπάρχει και μια ρήτρα διακοπής που έχει προσθεθεί στο πρωτόκολλο διακοπή της συμφωνίας εάν ένα από τα δύο μέρη παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για τη δυνατότητα διακοπής επίσης σε περίπτωση παραβιάσεων των κανόνων εργασίας βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Επίσης υπάρχουν ανησυχίες και στον τομέα αυτό, επίσης για πειρατικές δραστηριότητες που πλήττουν την αλληλεία και τους περιορισμούς που θέτουν στα νόμιμα αλληλευτικά σκάφη. Οι Σεϊχέλες είναι η μόνη κυβέρνηση, η μόνη που δέχεται να προσάγει στις δικαστικές αρχές ε, τους πειρατές και εδώ θα μνημονεύσω και την επιχείρηση Αταλάντη. Το 80% της αλίας του τόνου γίνεται από τα από τα γρηγρή και το υπόλοιπο από τα παραγαδιάρικα. Θα ήθελα εδώ να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πάρα πολύ περιοριστική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των αποθεμάτων, διμερείς συμφωνίες μεταξύ Σεϊχελών και τρίτων χωρών, που Μα δημιουργούν σημαντικέ ανησυχίε οι οποίες έχω συζητήσει και με την πρέσβυρα των Σιχελών στις Βρυξέλλες. το 2008 ο στόλο τη Ταϊβάν, τη Ιαπωνία, τη Κορέα και τη Κίνα, είχε ένα τεράστιο ποσοστό των, της αλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μόνο το 4% οι Ευρωπαίοι πλειοκτήτες δεν καταλαβαίνουν την αύξηση των ποσών που πρέπει να καταβάλουν, αυτό φαίνεται και από τη Νέα Συμφωνία, τα τέλη που καταβάλουν οι Ευρωπαίοι πλειοκτήτες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά υψηλά. Αυτό βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην μία ανανέωση ε, της συμφωνίας. Ναι, μπορούν, μπορούν να το καταβάλουν αυτό, ήθελα να πω, οι Ευρωπαίοι πλειοκτήτε, το ποσό αυτό. Η συμφωνία είναι σε γενικέ γραμμές αποτελεσματική, διότι ε, διασφαλίζει την παρουσία των ευρωπαϊκών σκαφών στην περιοχή, δίνει στις αιχέλες τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια υπεύθυνη βιώσιμη αλληλεία Οι επιστημονικές έρευνες μας δείχνουν ότι τα αποθέματα προστατεύονται, ότι σταθεροποιείται η ευρωπαϊκή αγορά κονσέρβα τόνου και αυτό βασίζεται εν μέρη και στην ύπαρξη αυτής της συμφωνίας. Νέες συμφωνίες συνεργασίες στα πλαίσια της αλληλείας ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στα πλαίσια μιας αλληλευτικής πολιτικής βιώσιμης και της υπεύθυνη εκμετάλλευση των αληφτικών αποθεμάτων της περιοχής. Αυτό βεβαίως δίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη Δημοκρατία των Σεχελών και στους πλειοκτήτες την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν την συμφωνία. Δεν βλέπω πολλούς ε, εδώ παρόντες αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν μείνει καλύτεροι. Περιμένω τα σχόλιά σας και σας ευχαριστώ για την μέχρι τώρα συμμετοχή σας. Κοιτάξτε, εκτό από ένα συνάδελφο, όλοι οι υπόλοιποι εδώ που έχουν είναι γυναίκες. Κυρία Μπλμπάου, Ευχαριστούμε κύριε Καντέκη για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Εγώ γενικά θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτή η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στη Μικτή Επιτροπή στην οποία γίνεται αναφορά σε άλλε συμφωνίες, να ζητήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και στην ενημέρωση, γιατί πρέπει να αναθεωρήσουμε τα έγγραφα. Ίσως ε, δεν είναι η καλύτερη διαδικασία για να εργαζόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο, όταν τα έγγραφα έρχονται πολύ αργά. Επίσης, ε, να ζητήσουμε να ελέγχουμε καλύτερα τα πολιετή, προγράμματα που εκπονούνται και να έχουμε και πρόσβαση στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ε, τώρα. Ακούσαμε τα αρνητικά στοιχεία που αναφέρετε, αλλά δεν θα τα επαναλάβω. Θέλω να πω ότι γενικά είναι σημαντική αυτή η συμφωνία για τον ε, ευρωπαϊκό στόλο της Ευρώπης. Έχουμε 70 σκάφη ε, και παραγαδιάρικα και γρηγρή τα 48 εργαλεία, τα υπόλοιπα παραγαδιόρικα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε τους 6.000 ε, τόνους ε, και είναι το ένα ε, τέταρτο μόνο του τόνου που αλλιεύεται εκεί ενώ το υπόλοιπο αλλιεύεται από σκάφη της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τα τελευταία έτη, λόγω των προβλημάτων της πειρατεία, η χρήση του πρωτοκόλλου και των πόρων που είχαμε μειώθηκε σημαντικά. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πέρα από την επιχειρήση Ατλαντίδα, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι δεν είχε σχεδιαστεί για να προστατεύσει τα λευτικά σκάφη η επιχείρηση αυτή. Αλλά χάρη στην κρίση που ανέκυψε με ε, την ε, κράτηση του σκάφους ε, που συζητήθηκε αυτό το θέμα και στο Κοινοβούλιο και εγκρίναμε στην επιχειρήση Ατλάντα να παρέχεται προστασία και στα ελευτικά σκάφη. Έτσι λοιπόν, ε, να επανέλθω να σας πω ότι τα ίδια τα σκάφη, τα γαλλικά σκάφη έχουν ε, στρατιωτικούς ε, επί του σκάφους και στα ισπανικά σκάφη υπάρχει προσωπικό προστασίας Θέλω λοιπόν να πω ότι πρόκειται για ένα είδο που θίγεται τα μάλα, αλλά και στο μέλλον θα θίγεται από αυτή την κατάσταση. Είναι καλό τα ευρωπαϊκά σκάφη να βρίσκονται εκεί, γιατί εμείς αποτελούμε την εγγύηση για μια υπεύθυνη και αηφόρο αλεία. Υπάρχουν λοιπόν παρατηρητές ε, σε όλα τα σκάφη που διορίζονται από την ίδια την κυβέρνηση των ΣΥΧΕΛΟΝ. Πιστεύω ότι λειτουργεί αρκετά καλά αυτό το σύστημα και φυσικά γνωρίζουμε και το ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα της δουλειάς μας εκεί, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις ΣΥΧΕΛΕΣ. Η δική μας ψήφος θα είναι θετική για την έγκριση της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ κυρία Λόβιν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφέρω δύο σημεία. Το ένα όσον αφορά την τομεακή περιφερειακή πολιτική σε αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα να ακούσω κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ Σεϊχέλων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μικτής Επιτροπής. Θα ήθελα να ξέρω πώς χρησιμοποιήθηκαν τα ποσά, σε ποια συγκεκριμένα προγράμματα της Επιτροπής. Δεύτερη ερώτηση. Η αλληλεία FAD. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα το γόνο του τόνου. Ε, πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις ε, πρακτικές. Σας έχει ενημερώσει η Επιτροπή. Πώς θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Πώς θα μειωθεί αυτή η δραστηριότητα και πώς θα μειώσουμε τα παραλιεύματα. Ο κύριος Κρόβατσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να παρατηρήσω πως ε, εμείς επιθυμούμε να υπάρχει ισότητα των φίλων ανδρογυναικών. Σε ό,τι φορά τώρα την ερώτησή μου, δεν ξέρω κατά πόσον θα πρέπει να την απευθύνω στον ε, εισηγητή ή ε, στην ε, Επιτροπή. Πώς από τα κονδύλια ε, εισπράττει η εισπράττει η σεισελ Μπάρια. Ευχαριστώ. Να πω πως η συμφωνία αυτή καταδεικνύει πως θα πρέπει να έχει μια εταιρική σχέση είναι μια συμφωνία που αποφέρει θετικά αποτελέσματα για την διατήρηση των πόρων Επίσης επηρεάζει τις θέσεις απασχόλησης ε, στις χώρες καταγωγής ε, και τις επιπτώσεις που έχει στην απασχόληση την Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα όπως αυτό της πειρατείας. Η συμφωνία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή η παρουσία μας ε, έχει ως ε, συνέπεια την ε, καταπολέμηση της παράνομης και λαθρέας αλίας. Ως εκ τούτου συμφωνούμε με την έκθεση του κ. Καντέκ, θα την υπερψηφίσουμε και η συμφωνία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα των όσων θα ακολουθήσουν για τα θέματα ενίσχυση ε, της ανάπτυξης, ε, προστασία των δικαιωμάτων κλπ. Κύριος Μπέρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Καντέκ που παρουσίασε με τρόπο ιδιαίτερα πλήρη τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας. Η κυρία Μπελέρα μίλησε για συμφωνία πρότυπο. Μας ικανοποιεί λοιπόν, είχαμε καλή συνεργασία με με τις Αιχέλες ε, την εφαρμογή του προηγούμενου πρωτοκόλλου και η τρέχουσα συμφωνία είναι μια συμφωνία που στηρίζεται σε υγιείς βάσεις. Έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμφίβολα τα ποσά σχετικά με την επιπτώση στον τομέα της απασχόλησης ε, μας το λένε, πρόκειται για χιλιάδες θέσεις εργασίας ε, τόσο στις ΕΧΕΛΕΣ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, είναι απολύτως ικανοποιητικά, καθησυχαστικά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σε ό,τι αφορά την διατήρηση των αλλιευμάτων στην περιοχή των ΣΕΙΧΕΛΟΝ η μεικτή επιτροπή που συνήλθε την 11η Φεβρουαρίου 2011 μας επέτρεψε να κάνουμε κάποια πρόοδο. Επανέρχομαι διότι είναι ένα θέμα που έθιξαν διάφοροι βουλευτές. Πώς έχει λοιπόν αυτή η κλαδική στήριξη, πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια αυτά. Υπήρχαν κάποια υπόλοιπα από το προηγούμενο πρωτόκολλο που μεταφέρθηκαν ε, σε έτη 2011 έως 2013. Για το 2011 φτάνουμε σε ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ με διάφορα μέτρα που παρουσιάζουν τρεις προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα βελτίωση της διαχείρισης της αερολίας τόσο της ε, βιομηχανικής όσο και της ε, αεραστεχνικής. Ε, αυτή είναι η πρώτη στην προτεραιότητα αυτού του τριετούς προγράμματος. Δεύτερος άξονας είναι οι υποδομές και εδώ υπάρχουν σημαντικά προγράμματα, σχέδια υποδομών, ιδιαίτερα η ανανέωση του λιμένα του για την αλία και η επέκταση του λιμένα για την βιομηχανική αλία αλλά και την τεχνική στήριξη για την συμφωνία αυτή και την οικοδόμηση ικανοτήτων. Τώρα, θα μπορέσουμε φυσικά να επανέλθουμε σε κάποιες λεπτομέρειες στις συμφωνίες αυτές. Έχουμε κάποιες ρήτρες ε, σύγχρονες θα έλεγα, έχουμε τις ε, ρήτρες ε, ανάκλησης σε περίπτωση μη στήριξη του κλάδου, είναι ρήτρες ναι, σύγχρονες γενιάς Κάτι ακόμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κατά πολέμηση της πειρατείας και κατά της παράνομης και λαθρέας και άναρχης αλίας. Να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την προσπάθεια που έχει καταβάλει ε, η κυβέρνηση των Σεϊχελών. Επίσης στηρίξαμε και ένα περιφερειακό πρόγραμμα εποπτείας του Ινδικού ωκεανού, το οποίο συμμετέχουν και οι Σεϊχέλες αλλά και πέντε ακόμα περιοχές, ε, μάλλον χώρες της περιοχής και που αποδίδει ικανοποιητικά σε όλη φορά την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας άναρχης ε, αλίας. Ε, η Σεχέλες είναι από τα πλέον δραστήρια μέρη για την προστασία στον Ινδικό ωκεανό. Τώρα, η ερώτηση για Λεβίν σχετικά με ορισμένες τεχνικές αλληλεία ε, που χρησιμοποιούνται και μπορεί να ε, αμφισβητηθούν συζητούνται στο Κολόμπο, στη Σρι Λάγκα, στο πλαίσιο της ε, οργάνωσης αλίας του ενδικού Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να εξετάσουμε, αλλά μόνο σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να απαντηθεί. Νομίζω πως ε, έδειξα τις περισσότερες, μάλλον όλες ερωτήσεις, ε, εκτός από το ποσοστό των εισοδημάτων ζυχελών ε, που προέρχονται από την συμφωνία. Δεν έχω τα στοιχεία υπόψη μου. Θα ενημερωθώ και θα σας τα αποστείλω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. για τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Σαφώς και δεν μπορεί αυτή η συμφωνία να είναι τέλεια. Σίγουρα όμως θα είναι παραδειγματική. Το λέω και το επαναλαμβάνω. Και πιστεύω θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο που οφείλεται κυρίως στην ε, ενεργό συμμετοχή των Σεϊχελών ή ιδιαίτερα μέσω κάποιων δράσεων που έχουν αναλάβει κατά της παράνομης λατρείας λίας, κατά της πειρατείας. Οι Σεϊχέλες όντες συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις και αυτό είναι σημαντικό για μας. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουμε πολύ προσεκτικοί. Η παράνομη λατρεία αναρχελία είναι κάτι που συνεχίζει και μας απασχολεί. Αν θέλετε να μου υποβάλλετε κάποια σχόλια, έχουμε βεβαίω επεξεργαστεί πολύ το κείμενο, αλλά αν έχετε κάτι που θέλετε να προσθέσετε, είμαι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ημερησία διάταξη για σήμερα το πρωί. Να σας ενημερώσω την επόμενη συνεδρίαση της 12 Απριλίου θα παρουσιάσει ο κ. την εκθεσή του και προβλέπεται να ψηφιστεί το Μάιο και να πάει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συνεδρίαση για σήμερα το πρωί. Έχετε κάποια ερώτηση διαφορετικά. κλείνουμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 3, ε, οπότε θα έχουμε και κλεισμένο των θυρών ανταλλαγή απόψε με εκπρόσωπο της Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ελίας με τις τρίτες χώρες και τις διαπραγματεύσεις. Λήξη της συνεδρίασης μέχρι τις 3.